Uh, dear Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Πρωί-πρωί εδώ είσαστε. Μετά από ολονύχτια ακρόαση, παρακολούθηση κλπ. Θεώρησα ότι ήταν μόνος μου στην συνεδρία της Επιτροπής Ήτρε. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Έχουμε πολύ σημαντικό θέμα να συζητήσουμε. Την ενεργειακή παινία. Ακρόαση. Now, may, Λοιπόν, έγκριση μερίσιας διάταξης. Άνευ σχολείου εγκρίνεται αμετάβλητη η μερίσια διάταξη. Δεν βλέπω να υπάρχει σχόλιο. Στο τέλος της συνεδριάσεως, πέμπτη δηλαδή, αύριο, 18 και 30 θα έχουμε τα διάφορα. Σας παρακαλώ λοιπόν να περιμένετε μέχρι τις 18 και 30 της Πέμπτης για να θέσετε ε, θέμα ή να δώσετε πληροφορίες. Ανακοινώσεις μου. Πολύ σημαντικό. Αύριο στις 9 θα γίνει ψηφοφορία για το σχέδιο εκθέσεως για τις δημιουργικές βιομηχανίες. Δική μας ιδέα μαζί με την Επιτροπή Πολιτισμού ε, κινούμαστε στον τομέα. Θα έχουμε κοινή συνεδρίαση, η ψηφοφορία στην Ήτρε θα ξεκινήσει στις 10. 10. Ξεκινάμε εμείς στις 9, ψηφίζουμε τη δημιουργική βιομηχανία μαζί με την Επιτροπή Πολιτισμού και μετά μένουμε στην ίδια αίθουσα. Και στις 10 έχουμε τη δική μας ψηφοφορία. Συνάδελφε Ρούμπικ, ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ήτρε, τον κύριο Μπούζεκ, και να τον ευχαριστήσω που κατάφερε να υπάρξει το χρονοδιάγραμμα για την ΣΤΟΑ και χαίρομαι που έχουμε εδώ πέρα μια σειρά από επιστήμονες που είναι στην ε, ε, συνεδρίαση της Επιτροπής μας θα μας παρακολουθήσουν για τρεις μέρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχαμε χθε τη μεγάλη ανοιχτή συνεδρίαση μαζί τους και έχουμε και εμπειρογνώμονες στα θέματα των τηλεπικοινωνιών. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους ε, βουλευτές για τρεις μέρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έρθουν σε επαφή με τους ε, εμπειρογνώμονες, τους επιστήμονες και για αυτή την πρωτοβουλία θέλω να σας ευχαριστήσω. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη συνεδρία τη Επιτροπή. Δεν ξέρω ακριβώ που καθέστε σε ποια θέση είσαστε. Μπορείτε να σηκώνετε το χέρι σα, παρακαλώ. Αν έχετε την καλοσύνη. Καλώ, καλώ. Σα ευχαριστώ που είσαστε εδώ στη συνεδρία τη Επιτροπή μα η δραστηριότητά σας ε, επίσης για τις προτάσεις στο Α και η παρουσία σας στη συνεδρίαση στο Α υπήρξε πάρα πολύ ε, ενεργός εκτές. Είχαμε πολύ φορτωμένη μέσα διάταξη. Ευχαριστώ συνάδελφε Πολ Ρούμπικ σαν πρόεδρος της στο Α οργανώσατε όλες τις ε, εκδηλώσεις. Άλλη ανακοινώση Δευτέρα 21 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο θα έχουμε κοινή συνεδρίαση Άγκρι Envy Ήτρε για την εφαρμογή Τη νέα ε, πολιτική Ευρωπαϊκή ενώσεω για τα δάση. Πολύ σημαντικό. Από τι 7 μέχρι τι 8 και 30. 7 με 8 και 30 στο Στρασβούργο. Δευτέρα 21 Νοεμβρίου. 7 με 8 και 30. Άγκρι, Ένβη, Ήτρε. Η στρατηγική, η δασική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πολύ σημαντικό θέμα και τις επιτροπέ από κοινού θα το συζητήσουμε. Πάμε στο εργαστήριό μα για την ενεργειακή παινία. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω όλου στο εργαστήριο αυτό για την ενεργειακή φτώχεια. Αυτή η ενεργειακή φτώχεια πραγματικά όλο και περισσότερο γίνεται θέμα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 50 με 125 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση απίστευτο κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν αυτή την ενεργειακή παινία. Υπάρχουν διάφορα αίτια όπως χαμηλό εισόδημα, υψηλή τιμή της ενέργειας, χαμηλή αποδοτικότητα η ενεργειακή αλλά υπάρχουν διάφορα αίτια. Αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Δεν υπάρχουν χρήματα για να πληρώνονται οι λογαριασμοί. Δεν έχει σημασία το αίτιο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αναμένεται ότι η μετάβαση προς μια οικονομία που δεν είναι ανθρακοβόρα μπορεί να ε, οδηγήσει και πολλούς άλλους ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα λόγω της αυξήσεως του κόστους για την μεταβατική περίοδο. Η Επιτροπή Ήτρε πάντα ασχολήθηκε με αυτό το θέμα στις εργασίες της αισθανόμαστε ότι έχουμε ευθύνη γι' αυτό. Να υπενθυμίσω ότι στο ψήφισμα του 2015 προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση ζήτησε το Κοινοβούλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει ανακοίνωση για την ενεργειακή παινία. Ορισμός, δείκτες για την ενεργειακή φτώχεια και να συνοδεύεται από σχέδιο δράσεως όσον αφορά την καταπολέμηση του φαινομένου. Τέλος, περιμένουμε προτάσεις λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε λύσεις για το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας. Η οδηγία η ενεργειακή αποδοτικότητα, η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων. Απόδοση κτηρίων σημαίνει ενεργειακή αποδοτικότητα επίσης και αναθεώρηση ε, για τους κανόνες περί σχεδιασμού των κτηρίων. Έχουμε πέντε νομοθετήματα για, ηλεκτρική ενέργεια, για το σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα μήνα. Και αυτά θα προταθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτό το πλαίσιο οργανώσαμε αυτό το εργαστήριο, όπου εμπειρογνώμονε θα συζητήσουν το θέμα από θεωρητικό επίπεδο, ακαδημαϊκό επίπεδο και θα παρουσιάσουν τα πορίσματα έρευνας που ανετέθη από την Επιτροπή Ήτρες Εμπειρογνώμονες. Επιτρέψτε μου λοιπόν να αναφερθώ σε συγκεκριμένα σημεία. Πρώτος ομιλητής. Α, θα δημοσιευτεί η παρουσίαση στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ήτρε και μετά συνοπτική έκθεση του εργαστηρίου θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Και να υπενθυμίσω στους ομιλητές ότι έχουν ένα τέταρτο στη διάθεσή τους για κάθε παρουσίαση. 15 λεπτά, όχι περισσότερα, σας παρακαλώ. Πρώτος ομιλητής. Σάσκα Πέτρουβα, που κάθεται δίπλα μου. για γεωγραφία στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Η δόκτωρ Πέτροβα θα αναφερθεί στην ενεργειακή παινία, το, το τοπίο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, από μια οπτική γωνία πανεπιστημιακή. Είναι πολύ καλά προετοιμασμένη διότι είναι καθηγήτρια στη Σχολή Περιβάλλοντος Παιδείας Ανάπτυξης και Διευθύντρια για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση στο Πανεπιστήμιο του Μάνσεστερ. Είναι και συντονίστρια των φατσερεύνες στο εργαστήριο για την αστυνομία ε, αντοχή, αν θέλετε, θεκτικότητα ε, στις, στο, όσον αφορά το περιβάλλον. Για την πόλη του Μάντσεστερ, όχι μόνο το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, εστιάζεται το έργο της επικοινότητας και τον, ε, το πλώς πλήττονται οι ντόπιοι από τη μετάβαση προς χαμηλές εκπομπές άνθρακα στις πόλεις και εξετάζει και τα θέματα του πόσο ευάλωτοι είναι οι άνθρωποι και ε, ποια είναι τα αποτελέσματα και επιτόσεις ενεργειακής αποδοτικότητας. Για το λόγο καθηγητρία, κυρία Πέτροβα. Ευχαριστώ, με ακούτε. Καλημέρα σε όλους και όλες. Μεγάλη χαρά είναι να είμαι εδώ μαζί σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οργανωτές που με προσκάλεσαν να συμμετάσχω και σε αυτό το εργαστήριο. Αυτή η συζήτηση καταδεικνύει και πάλι ότι η ενεργειακή ένδυα αποκτά όλο και μεγαλύτερη προσοχή μέσα στην ενεργειακή κοινότητα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει μπει στο λεξιλόγιο των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ήδη έχει, ολοκληρωθεί, έχει ενσωματωθεί η έννοια αυτή στο τρίτο ενεργειακό πακέτο και το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια. Η παρουσίασή μου θα εστιάσει στα σημαντικά επιστημονικά στοιχεία που συνδέονται με το θέμα της ενεργειακής ένδυας στην Ευρώπη. Στην αρχή της παρουσίασής μου θέλω να πω ότι η ενεργειακή ένδυα έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η έννοια με διαφορετικούς τρόπους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έλλειψη καυσίμων, η μη δυνατότητα να θερμαίνει κανείς το σπίτι του και η επισφάλεια στον τομέα της ενέργειας, όλα αυτά είναι απόψεις της ενεργειακής ένδυας. Αλλά η καλύτερη μορφή ορισμού ήταν από τον Μπρένταν Μπρόμαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος παρουσίασε ή Μπρόμαν παρουσίασε το θέμα αυτό ως την ανικανότητα ενός νοικοκυριού να έχει θέρμανση και άλλες ενεργειακές <clears throat> υπηρεσίες γιατί αυτό θα σήμαινε ότι πρέπει να δαπανίσει πάνω από 10% του εισοδήματό του νοικοκυριού για τέτοιες υπηρεσίες. Πιο πρόσφατότερα έχουμε συζητήσει τις ε, προτάσεις του οικονομολόγου Τζο Χιλ, ο οποίος εξετάζει τις συνέπειες ενός τέτοιου ορισμού. Αλλά πρότεινε ένα, νέο ορισμό μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι ο ορισμός του χαμηλού κόστους και του υψηλού εισοδήματος. Μα με μερικούς συναδέλφους, με τον κύριο Ποζορόφσκι και άλλους, Έχουμε επίσης προσπαθήσει να ορίσουμε με συνολικό τρόπο τι είναι η ενεργειακή ένδυα. Για μας και για το έργο μας, ο στόχος μας δεν είναι να περιγράψουμε μονάχα την σημερινή κατάσταση για τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά, <clears throat> αλλά να δούμε και κάποιες από τις αιτίε και τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν με την ενεργειακή ενδια ενός νοικοκυριού και τις συνθήκες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν το νοικοκυριό σε ενεργειακή ένδυα. Δεν είναι λοιπόν ένα στατικό φαινόμενο η ενεργειακή ένδυα. Μπορούν να μπουν αλλά μπορούν και να βγουν τα νοικοκυριά από την ενεργειακή ένδυα. Γι' αυτό ο δικό μα ορισμό είναι ότι είναι μια κατάσταση ή μάλλον μια, ένας συνδυασμός καταστάσεων που μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους να μπει ένα νοικοκυριό σε ενεργειακή ένδυα, κάτι το οποίο σημαίνει το νοικοκυριό δεν μπορεί να έχει μια υλική δυνατότητα να έχει τις υπηρεσίες ενέργειας που είναι κοινωνικά αποδεκτές. Πολλοί ακαδημαϊκοί έχουν πει ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει κοινό ευρωπαϊκό ορισμό για την ενεργειακή ενδιά. Άλλοι έχουν αντίθετη γνώμη. Ο Χάρι Τόμσον και άλλοι συνάδελφοι έχουν υπογραμμίσει το γεγονό ότι μια κοινή ενεργειακή ένας κοινός ενεργειακός ορισμός της ένδυας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αυξήσει την αναγνώριση και την πολιτική ορατότητα του προγράμματος στην Ευρώπη, αλλά μπορεί να επιλύσει και κάποια από την τερμι... ορολογιακή ε, σύγχυση, γιατί μερικές φορές έχουμε διαφορετική αντίληψη της ενεργειακής ένδυας και μπορεί να δημιουργήσει και πολυ σε συνέργειες σε επίπεδο πολιτικής με το να συνδέσει διάφορους τομείς. Κοινωνική πολιτική, βιομηχανία, υγειονομική πολιτική και καθαρά ενεργειακές πολιτικές σε ό,τι αφορά την αγορά ηλεκτρισμού κτλ. Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι όμως έχουν στραφεί εναντίον ενός κοινού ορισμού, γιατί κατά την άποψή τους ένας κοινός ορισμός μπορεί να ισοπεδώσει τις ιδιαίτερες γεωγραφικές καταστάσεις. Παραγωγή χάρη διαφορετικές κοινωνικο-οικονομικές καταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολιτικές ε, συγκυρίες και διαφορετικές ε, περιφερειακές καταστάσεις που μπορεί να υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να καταλάβουμε από πού προέρχεται η ενεργειακή ένδυα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι απαραίτητη. Παραδοσιακά η επιστημονική έρευνα έχει εντοπίσει τρεις κερίους παράγοντες, μεταξύ των οποίων το τίμημα της ενεργείας, η μείωση του εισοδήματος των οικοκυριών και η έλλειψη ενεργειακής αποδοτικότητος στα σπίτια που μένει ένα οικοκυριό. Αυτό είναι λοιπόν το τρίγωνο των πολιτικών και των κινδύνων που εξηγεί τη μορφή της ενεργειακής ένδυσης. Αλλά πιο πρόσφατα έχει τονιστεί η αποτελεσματικότητα στη χρήση της ενέργειας ως ένας κέριος παράγων για την αποτροπή της ενεργειακής ένδυας γιατί οδηγεί σε μεγαλύτερη ε, άνεση στα σπίτια από θερμική άποψη και από την άποψη της αποτροπής της υγρασίας. Επομένως βρίσκεται στην τομή της ε, σχέσης εισοδήματος, τιμών και ενεργειακής απόδοσης. Επομένως είναι μια μορφή υλικής αποστέρησης η οποία είναι κάτι περισσότερο από την απλή εισοδηματική ένδυα. Είναι μια πιο υλικότερη λοιπόν μορφή αποστέρησης για τα νοικοκυριά. Ακόμα και νοικοκυριά που έχουν υψηλές ανάγκες σε ενέργεια με παιδιά, με ηλικιωμένους κτλ. έχουν δείξει να είναι πιο ευάλωτα στην ενεργειακή ένδια. Είναι χρήσιμο λοιπόν να έχουμε πιο ευέλικτα συστήματα θέρμανσης τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια πιο προσβάσιμη οικονομικά ή τεχνικά πιο κατάλληλη μορφή παροχής ενεργειακών υπηρεσιών ώστε να ξεπεραστεί η ενεργειακή ενδια. Είναι απαραίτητο λοιπόν να λάβουμε υπόψη και τα θέματα της υγείας. Ξέρουμε λοιπόν ότι στον τομέα των νοικιαζομένων σπίτιων μπορεί να υπάρχουν μεγαλύτεροι κίνδυνοι για αυτούς οι οποίοι μένουν εκεί πέρα να γίνουν ενεργειακά φτωχοί. Ένα κατ' ότι δεν έχουμε ένα κοινό για το τι είναι η ενεργειακή ένδυα, είναι δύσκολο να ποσοτικοποιήσουμε την έκταση αυτού του φαινομένου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ συχνά οι ερευνητές χρησιμοποιούν τα στοιχεία της Eurostat που αφορούν το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης και επίσης το, την έρευνα για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Αλλά Αυτές οι έρευνες περιλαμβάνουν διαφορετικές μεταβλητές και επομένως επί τη βάση των μεταβλητών που επιλέγουν οι ερευνητές καταλήγουμε σε διαφορετικά στοιχεία για την ενεργειακή ένδια. Υπολογίζεται όμως η ένδια αυτή να καλύπτει από 50 ως 160 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονό ότι υπάρχει αυτό το χάσμα ενεργειακή ένδυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο είναι τεκμηριωμένο στην επιστημονική φιλολογία. Δείχνει ότι το φαινόμενο αυτό βρίσκεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίω στην Ανατολική και Νότια Ευρώπη. υπάρχουν διαφορετικοί δείκτες και διαφορετικοί ενδείκτες που καταδεικνύουν ότι τα επίπεδα ενεργειακής ένδυας είναι υψηλότερα στη Βουλγαρία, στην Κύπρο και στη Ρουμανία. Πολλές ακαδημαϊκές μελέτες έχουν υπογραμμίσει υψηλά επίπεδα ενεργειακής ένδυας σε πρώην σοσιαλιστικές ε, χώρες έχουν να κάνουν με την αύξηση του τιμήματος ενέργειας μετά τη φιλελευθερωποίηση της αγοράς ενέργειας. η έκθεση Μποζαρόφσκι και Θηράδο Ερέρο έδειξαν ότι στην Πολωνία έχουν αυξηθεί οι τιμές κατά 33%, 22% στην Τσεχική Δημοκρατία και 69% στην Ουγγαρία μεταξύ 2006 και 2011. Τα επίπεδα ενεργειακής έργειας ήταν επίσης πάρα πολύ ψηλά σε χώρες της Νότιας Ευρώπης λόγω επειδή δεν υπάρχουν αποτελεσματικές ε, κατοικίε σε ενεργειακό επίπεδο. Οι χώρες της Μεσογείου επίσης, νότιας Μεσογείου, έχουν το πρόβλημα της ε, ψήξης των ε, οικειών τους το καλοκαίρι. Έχει λοιπόν υπολογιστεί ότι περίπου το 1 τρίτο αυτών οι οποίοι απάντησαν στα, 18, στα 8 κρατημέλη που βρίσκονται στη Μεσόγειο δεν ήταν σε θέση να κρατήσουν τα σπίτια τους σε μια αποτελεσματική και άνετη θερμοκρασία και να ψύχουν τα σπίτια τους το καλοκαίρι. Το καθεστώς λιτότητας στην Ελλάδα επίσης έχει επηρεάσει και το επίπεδο ενεργειακής ένδυας στην ταλαιπωρημένη αυτή χώρα. Κάτι που μπορεί να είναι επίσης σημαντικό για την έκταση της ενεργειακής ένδειας είναι οι ενεργειακές μεταβάσεις, όπως είπε πολύ σωστό ο κ. Μπουζαρόφσκι. Αυτές οι ενεργειακές μεταβάσεις χαιρετίζονται από την απανθρακοποίηση των ενεργειακών συστημάτων. Είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να επηρεάσει κυρίως νοικοκυριά χαμηλού ε, εισοδήματος όταν η απανθρακοποίηση, οι επενδύσεις στις ε, ε ανανεώσιμες ενέργειες μετακυλίονται στον καταναλωτή με αυξημένα τιμήματα ενέργειας η φορολογία του δίζελ και της βενζίνης και σε μικρότερο βαθμό του φυσικού αερίου είναι λιγότερο αρνητικές για τους στοχούς, αλλά η φορολογία του ηλεκτρισμού είναι πιο αρνητική για τα φτωχά νοικοκυρία, όπως έχει δείξει μια σειρά από μελέτες. Ακόμα όμως, πολλοί ακαδημαϊκοί μελετητές υποστηρίζουν το επιχείρημα ότι οι οικουμενικές επιδοτήσεις για την ενέργεια δεν είναι ένα αποτελεσματικό αναδιανεμητικό εργαλείο γιατί τα πιο πλούσια νοικοκύρια κατανάλωνουν πιο πολύ ενέργεια από ό,τι τα φτωχά. Γι' αυτό το... η στήριξη του εισοδήματο με τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική. Άλλες έμεσες μέθοδοι μπορεί να περιλαμβάνουν την υποστήριξη των δημόσιων ε, μεταφορών και αναβάθμιση των σπιτιών. Επίσης έχει αναφερθεί ότι η μετάβαση σε οικονομία χαμηλού ανθρώπους μπορεί να είναι πιο δίκαια αν ε, χρηματοδοτείται από την φορολογία εισοδήματος. Και έχω τώρα και μία σύνοψη των κύριων σημείων που ανέφερα, <clears throat> γιατί δεν ξέρω τι έχω ξεπεράσει το χρόνο, μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτά τα ε, συμπεράσματα και στο τέλος της ε, παρουσίασής μου θα σας πω ότι έχω και μία βιβλιογραφία, εάν κάποιοι από εσά ενδιαφέρονται να πάρουν περισσότερες πληροφορίες και επίσης θα ήθελα να σας αναφέρω ότι έχουμε ένα σχέδιο το οποίο αφορά σε μερικές από τις πιο ε, ευ... χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Πολωνία Βρισκόμαστε σε τρεις πόλεις και έχουμε κάνει και μελέτες σε άλλες ε, χώρες και πόλεις για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία. Ο επόμενος ομιλητής μας είναι ο κύριος Μπενιαμίν Γκράινερ, ο οποίος είναι ερευνητή στο Ινστιτούτο ΕΚΟ του Βερολίνου. Είναι ένας ε, εκπαιδευμένος ε, επιστήμονας πολιτικός που έχει ασχοληθεί πολύ με την βιώσιμη ανάπτυξη. Έχει εμπειρία σε θέματα πολιτικής, οικονομικών, κλιματικής αλλαγής, προσαρμογής και διεθνούς ανάπτυξης και όσον αφορά τις τεχνολογικές μεταβάσεις, κάτι στο οποίο αναφέρθηκε και η κυρία Πέτροσκα. Δουλεύει στο Ινστιτούτο αυτό στο Βερολίνο από το 2014. Έχει εργαστεί στην, ε, στο σχεδιασμό αξιολογήσεων, στην ε, επιθεώρηση και αξιολόγηση πολιτικών τόσο στη Γερμανία όσο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρίε και κύριοι. Μεγάλη τιμή για μένα που απευθύνομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Θα σας παρουσιάσω μια μικρή μελέτη που κάναμε πέρυσι και που μας ανέθεσε η Επιτροπή Ήτρε σχετικά με την κατάσταση της ενεργειακής ένδυας σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Ποιες είναι οι προδιαγραφές και κάναμε και μια αξιολόγηση των δυσκολιών που διαπιστώνουμε όσον αφορά τις πολιτικές των χωρών μελών σχετικά με την ενεργειακή ένδυα. Λοιπόν, τι κάναμε. Κάναμε μία μελέτη ερευνητική, δηλαδή προσπαθήσαμε να συλλέξουμε στοιχεία, δεδομένα και να δούμε αν υπάρχει κάποιο μοντέλο που ακολουθείται. Εμείς δεν ελέγξαμε τις υποθέσεις εργασίας, απλώς καταγράψαμε την εικόνα του τι συμβαίνει στην ε, χώρα, στις χώρες μέλη. Είχαμε, συγκεντρώσαμε λοιπόν μελέτες από διάφορες χώρες, μιλήσαμε με εμπειρογνώμονες και με ερευνητέ από τις διάφορες χώρες μέλη. Η ενεργειακή ένδια λοιπόν είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπω είπε και η δεν θα μπω σε λεπτομέρειε. Αλλά όπω βλέπετε είναι ένα πρόβλημα σε πολλέ χώρε μέλη. Δεν περιορίζεται στι πιο φτωχέ χώρε μέλη, μόνο στο βορρά, μόνο στην είτε, στο νότο. Η Ισπανία και η Ελλάδα πλήττονται εξίσου, όπω και άλλε χώρε του βορρά. Δεν μπορούσαμε βέβαια να μπούμε σε λεπτομέρειε σε όλες τις χώρες μέλη. Επιλέξαμε με γεωγραφική διαφοροποίηση βορρά-νότου, με οικονομική διαφοροποίηση υψηλών εισοδημάτων και χαμηλών εισοδημάτων και συγκρίναμε ευρωπαϊκές χώρες των 15 και χώρες μετά την ένταξη του 2004 διαπιστώσαμε τα ότι οι τιμές της ενέργειας αυξάνουν σε όλες τις χώρες μέλη. Και αυτό είναι πρόβλημα. Οδηγεί σε ενεργειακή ένδια και θα οδηγεί και στο μέλλον. Έχει να κάνει με μακροοικονομικούς δείκτες. Σας είπα ότι δεν είναι οι πιο φτωχές χώρες που υποφέρουν από ενεργειακή ένδια. Είναι κάτι που αναγνωρίζει το πρόβλημα σε όλες τις χώρες μέλη. Υπάρχει πάντα στην ε, ατζέντα των χωρών μελών, συζητιέται και μερικές φορές αντιμετωπίζεται με κοινωνικές πολιτικές. Αλλά θα έρθω σε αυτό αργότερα. Οι ορισμοί πολιτικοί διαφέρουν και διαφέρουν και τα στοιχεία που έχουμε. Τώρα θα έρθω σε λεπτομέρειες σχετικά με διάφορες χώρες όπου ερευνήσαμε την κατάσταση. Η Ιρλανδία για παράδειγμα είναι μια χώρα δυτική, όμως έχει πολύ ενεργειακή ένδια, 20% περίπου και οπολογίζεται αυτό βάσει του κόσμου που θα πάνε κάτω από 10% και τις ενεργειακές του ανάγκες. Η ποιότητα των κτηρίων δεν είναι αρκετά καλή και στην Ιρλανδία υπάρχουν πάρα μεγάλες απαιτήσει για θέρμανση. Υπάρχουν διάφορες πολιτικές. Υπάρχει μια πολιτική που είναι η βελτίωση των κτηρίων, να είναι πιο αποδοτικά ενεργειακά και υπάρχει και χρηματοδότηση του ενεργειακού κόστους με προγράμματα για βελτίωση των κτηρίων και για επιδόματα. Επιδόματα για τον λογαριασμό ενέργειας που φτάνει στα νοικοκυριά ή για εξοικονόμηση πολλές φορές συγκεντρώνονται οι ανάγκες και αγοράζουν ε, πετρέλαιο τα νοικοκυριά πιο φτηνά όταν χοντρικά αγοράζουν πολύ μαζί. Η δεύτερη περίπτωση που εξετάσαμε ήταν η Γαλλία, η οποία ορίζει με ενδιαφέροντα τρόπο την ενεργειακή φτώχεια, όχι τόσο διαφορετικά από ό,τι ανέφερε η κυρία Πέτρο, πάντα είναι το 10% το όριο, αλλά η ενέργεια ορίζεται σαν ένα βασικό αγαθό στη Γαλλία άρα χρειάζονται και δικές πολιτικές. Οι εταιρείε κοινή ωφέλεια δεν μπορούν να κόψουν ε, την παροχή, για παράδειγμα. 3,5 εκατομμύρια νοικοκυριά στη Γαλλία βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία. Τώρα η Γαλλία βασίζεται κυρίως σε κοινωνικές ε, παροχές για τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα. Έχει και προγράμματα για βελτίωση των κτηρίων και με τις ενεργειακές εταιρείες που βοηθούν τον κόσμο να βελτιώσει την μόνωση στα σπίτια του. «50.000 κτίρια ανακοινήστηκαν με αυτό το τρόπο, ενώ πρόκειται για 3,5 εκατομμύρια νοικοκυριά. Δύσκολη περίπτωση. Α δούμε τη Βουλγαρία τώρα. Όπω είπε και η κυρία Πετρόβα, στι χώρε Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη δεν υπάρχει ενεργειακή πολιτική, δεν αποτελεί εξαίρεση η Βουλγαρία. Έχουν πολύ παλιά κτίρια και 50% του πληθυσμού κινδυνεύει γενικά από ένδια. Άρα και από ενεργειακή ένδια. Με προβλήματα στην υγεία, πρόωρους και κλπ. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό στη Βουλγαρία. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε στοιχεία για τα κτίρια στην Βουλγαρία και για τον κόσμο γενικά. Και είναι δύσκολο να προσφύγω σε πηγέ χρηματοδότηση στα νοικοκυριά. Υπάρχει βέβαια κοινωνική πολιτική που καλύπτει τη θέρμανση στη Βουλγαρία. Αλλά είναι για ένα δωμάτιο το χειμώνα να θερμαίνεται. Είναι τα πολύ βασικά και η βελτίωση των κτηρίων δεν είναι απαραίτητα για την ε, ενεργειακή βελτίωση. Τέλος έχουμε το Ηνωμένο Βασίλειο. Η συζήτηση για την ενεργειακή ένδια γίνεται από τη δεκαετία του 80 εκεί. Το ενδιαφέρον στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι λάζουν τους δείκτες. Έχουν μια πολύ περίπλοκη μεθοδολογία, η οποία βασίζεται στο κόστος που πληρώνει ο κόσμος και σε ένα υποθετικό μοντέλο κόστους, λαμβάνοντας υπόψη τα κτίρια, τις ενεργειακές ανάγκες και διαπιστώνουν πόσο θα έπρεπε να πληρώνουν οι άνθρωποι αυτοί για να θερμαίνουν τα σπίτια τους ικανοποιητικά. Έχουν βέβαια κάποια προγράμματα, αλλά η μεθοδολογία αυτή είναι πρόβλημα. Και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν δίνει πολλά επιδόματα αλλά είναι και τοπικές αρχές, η Βόρεια Ιρλανδία, η Ουαλία και τα λοιπά, που έχουν τα δικά τους επιμέρους προβλήματα. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο υπάρχουν υποχρεώσεις για τις ενεργειακές εταιρείε που πρέπει να βελτιώνουν τα μέτρα, να υπάρχει περιορισμό στι τιμέ. επίσης. Και το 2017 θα υπάρξουν παρετέρω μέτρα που θα εφαρμοστούν. Λοιπόν, ποιο είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών αυτών. Υπάρχει μια προσέγγιση τριών βημάτων. Το πρώτο βήμα είναι να ορίσουμε τι είναι, ποιος θεωρείται ότι υποφέρει από ενεργειακή ένδια. Το δεύτερο αποτελεί μέρος της ε, εφαρμογής, δηλαδή να εντοπίσουμε ακριβώς ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισμό αυτό. Και το τρίτο στάδιο είναι η εφαρμογή. Δηλαδή πώς θα βελτιώσουμε την κατάσταση των ανθρώπων αυτών. Βοηθάνε οι πολιτικές που έχουν μέχρι τώρα εφαρμοστεί ή όχι. Οι δυσκολίε είναι εξή. Πρώτα απ' όλα για το πρώτο στάδιο. Πώς δηλαδή ορίζεται η ενεργειακή ένδια. Η αρχή της δαπάνης για την ενέργεια είναι κάτι απλό. Αν είναι πάνω από 10% εντάξει, αν κάτω από 10% υποφέρει από ενεργειακή ένδυα. Οι άνθρωποι, και αυτό είναι πρόβλημα στην Ισπανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν προβλήματα υγείας ε, πολλοί λόγω προβλημάτων να πληρώσουν ε, για την ενέργεια, αλλά παρόλα αυτά δεν εμπίπτουν στον ορισμό. Η δεύτερη περίπτωση είναι τα χαμηλά εισοδήματα και το υψηλό κόστος. Είναι κάτι πιο περίπλοκο να υπολογιστεί. χρειάζονται πολλά στοιχεία για τα κτίρια και στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα που γίνονται προσπάθειες για να συλλέξει στοιχεία η κυβέρνηση, παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκτιμηθούν τα στοιχεία αυτά. Και τέλος δεν υπάρχει ένας πραγματικός ορισμός για την ενέργεια. Αν κάποιος παίρνει επιδόματα στην ε, Γερμανία για τη θέρμανση, αυτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητα υποφέρει από ενεργειακή ένδια το άτομο. Οπότε για να καταλήξει κανείς σε πολιτική πρέπει να τα συνδυάσει όλα αυτά πολύ καλά. Το χαμηλό εισόδημα δεν σημαίνει απαραίτητα και ενέργεια και ένδια. Εδώ υπάρχει το κομμάτι αυτό που βλέπετε που είναι κοινό στους δύο κύκλους. Αυτό μας ενδιαφέρει. Τελικά τι καλύπτουμε, ποιον από τους δύο κύκλους καλύπτουμε. Α δούμε τώρα τον εντοπισμό των νοικοκυριών που υποφέρουν από ενεργειακή ένδια. Ο καθηγητής, τον οποίο αναφέρθηκε προηγουμένω και η κυρία Περκοβά, έχει πει ότι το 1 τέταρτο των χρημάτων πηγαίνουν στον κόσμο που υποφέρει από ενεργειακή ένδια. Άρα λοιπόν είναι πρόβλημα εντοπισμό των οικοκυριών αυτών. Δεν υπάρχουν λεπτομερεί στοιχεία είναι δύσκολο να αποκτήσουμε τα στοιχεία, να τα δημοσιεύσουμε και να βασίσουμε τις πολιτικές μας πάνω σε αυτό. Και έπειτα υπάρχει και το στίγμα για αυτούς τους ανθρώπους, που είναι μεγάλο πρόβλημα και α μην το περιμένουμε. Δηλαδή και αυτοί που παίρνουν επιδόματα ε, αισθάνονται άσχημα και πολλές φορές διστάζουν να ζητήσουν βοήθεια. Θετική εμπειρία έχουμε στη Γαλλία για παράδειγμα, όπου τα επιδόματα αυτά τα δίνει η τοπική αυτοδίκηση. Οπότε είναι πιο εύκολο να εντοπίσει τα νοικοκυριά που έχουν πραγματικά ανάγκη, γιατί γνωρίζουν τους γειτονέ τους, γιατί γνωρίζουν τις ανάγκες και στη Γαλλία είναι πολύ αποτελεσματικό αυτό το σύστημα. Συνέπεια τώρα των δυσκολιών αυτών βλέπετε εδώ σε αυτό το πίνακα. Είναι βέβαια κάπως υποκειμενική αυτή η αξιολόγηση, ομολογώ, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι να, εδώ πάνω βλέπετε πολύ πράσινο, που σημαίνει ότι είναι στόχος η αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδυας σε αυτές τις χώρες. Μετά βλέπετε όλο και λιγότερο πράσινο όσο κατεβαίνουμε για τον εντοπισμό και για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών. Και κάτω-κάτω βλέπετε σκούρο πράσινο, γιατί σε αυτές τις χώρες βοηθούνται οι άνθρωποι να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, αλλά δεν αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές το βασικό πρόβλημα που είναι το χαμηλό εισόδημα και η χαμηλή απόδοση, ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Είναι πράγματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται. Χρειάζονται πολλά χρήματα. 300 εκατομμύρια στη Γαλλία για το καλύτερη στέγαση, αυτό το πρόγραμμα της Γαλλίας. Ας δούμε τώρα τα υπέρ και τα κατά των διάφορων πολιτικών. Υπάρχουν οι κοινωνικέ τιμέ ηλεκτρισμού και ενέργεια. Στην Ελλάδα και την Ισπανία εμφανίστηκε αυτό το μέτρο και ήταν θετικό. Ε, βοηθήθηκε ο κόσμο, αλλά δεν αντιμετωπίστηκαν οι ρίζε του κακού. Πολλοί βέβαια στην Ελλάδα ε, κινδύνευσαν και υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη πίεση στου πάροχου ενέργεια για να χαμηλώσουν τις τιμές τους. Αυτοί όμως μετά δυσκολεύτηκαν να πληρώνουν του δικού του λογαριασμού και ούτω καθεξής. Άρα είναι ένας οικονομικός φαύλος κύκλος. Η δεύτερη πολιτική είναι η στήριξη της ε, ανακαίνησης των κτηρίων στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι ένα καλό μέτρο γιατί αντιμετωπίζει την πηγή της ενεργειακής ένδυας. Ανακαινίζονται σπίτια και ο κόσμος που ρωτήθηκε είπε ότι βελτιώθηκε η κατάστασή τους, ότι δεν νιώθουν πια να κρυώνουν στα σπίτια τους το χειμώνα. Αλλά χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα ένα τέτοιο μέτρο και πρέπει τα κονδύλια αυτά να δοθούν εκεί που χρειάζεται. Είδαμε ότι η Βουλγαρία δυσκολεύεται να βρει χρήματα για την αντίστοιχη χρηματοδότηση. Πάντως είναι η μόνη πραγματική λύση που μακροπρόθεσμα φέρνει αποτελέσματα. Έπειτα η χαμηλή ενεργειακή απόδοση των κτηρίων ε, δεν σημαίνει απαραίτητα και ενεργειακή ένδια. Αν μιλάμε για ενεργειακή ένδυα λοιπόν, πολλοί οι οποίοι ζουν σε κτίρια με κακή ενεργειακή απόδοση μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Και το τρίτο είδος πολιτικών είναι τα επιδόματα για την ενέργεια σε νοικοκυριά χαμηλών εισοδημάτων. Έχει βέβαια μικρό διοικητικό άκθος αυτό, αλλά πάλι δεν αντιμετωπίζεται η πραγματική πηγή της ενεργειακής ένδυας, ούτε των χαμηλών εισοδημάτων και της απόδοσης των κτηρίων. Όταν έχετε τόσα πολλά νοικοκυριά που υποφέρουν από ενεργειακή ένδυα όπως στη Βουλγαρία, το να εντοπιστούν οι άνθρωποι δεν είναι τόσο πολύ πρόβλημα γιατί πληρώνεις γενικά ένα επίδομα για την ενεργειακή ένδυα και καλύπτεις όλο αυτό το κόσμο. Δεν πάνε τόσο χαμένα τα χρήματά σου, αλλά σε άλλες χώρες είναι αλλιώς. Οι προκλήσεις είναι και οι δυσκολίες. Η έλλειψη στοιχείων για την ποιότητα των κτηρίων, ο εντοπισμός των ε, νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να πληρώσουν τους ναριακούς τους λογαριασμούς, η επαρκής χρηματοδότηση και η εφαρμογή μακροπρόθεσμων λύσεων. Τι μπορούμε να κάνουμε. Θα έπρεπε όπως κάνει και το Ινστιτούτο μας, να συλλέγουμε στοιχεία. Αλλά δυστυχώς δεν είναι λεπτομερή για όλες τις χώρες μέλη. Θα έπρεπε επίσης να υπάρξουν περισσότεροι δίωδοι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε λύσεις. Στη Γερμανία υπάρχει δυσκολία στέγασης, γιατί δεν υπάρχουν αρκετά κτίρια για στέγαση. Η ενεργειακή ένδια, έτσι καλλιώς, είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και ευχαρίστω να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. τόσο ομιλητής. Ο κύριος Σέρτζιο Ουγκάρτε, διευθυντής και σύμβουλος. Έχει πάνω από 25 χρόνια υπηρεσία στον τομέα της παροχής συμβουλών για τη συναλλαγή της ενεργικής πολιτικής και στρατηγικές για διάφορους πελάτες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ευρώπη και σε άλλες υπήρους. Είναι δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο. Έχει τεράστια γνώση όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα, στρατηγικές για τις χαμηλές εκπομπές άνθρακα στη βιομηχανία, μελλοντικές ενεργειακές, ε, ανάγκες ηλεκτρική ενέργεια, ενεργειακές στρατηγικές κλπ ανάπτυξη του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νέος σχεδιασμός του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορούμε να πούμε με αυτή τη βάσεις ότι έτσι καταπολεμούμε και την ε, ενεργειακή ένδια. Ε, λαμβάνουμε υπόψη αυτό το στοιχείο στον ενεργειακό σχεδιασμό. Θα θέλαμε τις συμβουλές σας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους, ε, λέει ο κύριος Σουγκάρτε. Με τα χαράς να παρουσιάσω τα απορίσματα της μελέτης που ανετέθη από την Επιτροπή σε εμά όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα για νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα. Αυτή η μελέτη δίνει με συνέχεια στην μελέτη που έκαναν οι συνάδελφοι εδώ του Ινστιτούτου που εξέτασε ήδη σφαιρικά τις κοινωνικές πολιτικές και τις πολιτικές εν γέννη στην ε, Ευρώπη αυτή η μελέτη εδράζεται κατά πολύ στις γνώσεις και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν ο σημαντικούς επιστήμονες στην Ευρώπη, όπως ε, η δόκτωρ Πεντρόβα και άλλοι συνάδελφοι έκαναν τέτοιες μελέτες όσον αφορά τον καθορισμό της ενεργικής ένδυας και την ανάλυση των σχετικών κινδύνων. Ξεκινώντας λοιπόν. Γνωρίζουμε ήδη τον κίνδυνο της ενεργειακής ένδυας. Έχουμε κάποια στοιχεία όσον αφορά τον αριθμό των ανθρώπων που υποφέρει αυτό το φαινόμενο Ξέρουμε ότι τα ριζικά αίτια δεν είναι μόνο το χαμηλό εισόδημα, αλλά και το ποσό της ενέργειας που χρησιμοποιεί ένα νοικοκυριό. Αν νοικοκυριό δεν έχει ενεργειακή αποδοτικότητα, χρησιμοποιεί περισσότερη ενέργεια από ένα άλλο νοικοκυριό. Και αν επιπλέον οι κάτοικοι του νοικοκυριού αυτού έχουν χαμηλό εισόδημα, οι ένικοι, δεν μπορούν να πληρώσουν αυτό τον μεγάλο λογαριασμό. Ε, λόγω που προξενείται από τη μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Άρα η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική μεταβλητή στην εξίσωση της ενεργειακής ενδίας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την ενεργειακή αποδοτικότητα για να μειώσουμε το κόστος που αντιμετωπίζει ένα νοικοκυριό με χαμηλό εισόδημα για την ενέργεια. Αυτό και όχι μόνο να καθορίσουμε τις κοινωνικές πολιτικές που θα διοχετεύουν δημόσιο χρήμα μέσω επιδοτήσεων για να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά να περάσουν το χειμώνα και να έχουν μια κάποια ελάχιστη άνεση. Πού εστιαζόμεθα λοιπόν επί ενεργειακής αποδοτικότητας σε νοικοκυριά. Ποιες είναι οι συνέπειες, αυτό είναι το πρώτο ερώτημα, της ενεργειακής αποδοτικότητας για τα φτωχά νοικοκυριά. Καταρχάς, ε, το περιβάλλον επηρεάζεται. Ε, βοηθάμε το περιβάλλον μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας. Αυτός δεν είναι ο πιο σημαντικός αντίκτυπος για την οικοκυριά, αλλά οι κοινωνικές συνέπειες, οι οικονομικές συνέπειες. Ε, πέρα της μειώσεως των εκπομπών, μπορούμε να βοηθήσουμε τη βελτίωση υγείας των ενίκων των οικοκυριών, μειώνοντας επίσης και το λογαριασμό πληρών για την υγεία τα κράτη. Μπορούμε να βοηθήσουμε τους τα κράτη να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις απασχόλησης, ε, να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, κυρίως ε, για τους νέους και τα παιδιά. Υπάρχει ποικιλία λοιπόν κοινωνικών ε, ωφελιών που απορρέουν από την ενεργειακή αποδοτικότητα. Λοιπόν, πέραν της πληρωμής ή μη πληρωμής του λογαριασμού, που καλύπτεται από κοινωνικές πολιτικές, τα κοινωνικά ευεργετήματα από την ειδική αποδοτικότητα ε, είναι πολύ σημαντική συνιστόσα και πρέπει να εστιαστούμε από αυτού. Μετά να ρωτήσουμε το εξή. Ποιοι είναι οι φραγμοί όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα, αν είναι τόσο σαφές και λογικό να την επιδιώκουμε, γιατί υπάρχουν ε, τόσα νοικοκυριά με χαμηλή ενεργειακή αποδοτικότητα. Ποια είναι τα προβλήματα, φραγμοί για την νοικοκυριά. Πρώτα απ' όλα έλλειψη πληροφόρησης δεν έχει ο κόσμος τις κατάλληλες πληροφορίες. Πώς να εξοικονομήσει ενέργεια. Οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες των ανθρώπων. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει έλλειψη γνώσης που συνδυάζεται και με χαμηλό εισόδημα και αυτός ο συνδυασμός περιπλέκει την κατάσταση. Δεν είναι γενικό αυτό. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ανατολική Ευρώπη άνθρωποι με πολύ καλή εκπαίδευση δεν μπορούν να πληρώσουν τον λογαριασμό τους διότι έχουν καταναλώ πολύ ενέργεια λόγω έλλειψης μόνωση στα σπίτια. Άλλο είδους πρόβλημα φραγμή. Δεν υπάρχει πρόσβαση στο χρήμα. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν πώς να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους αλλά δεν έχουν τα χρήματα να επενδύσουν για να το πετύχουν αυτό. Ακόμα και αν γνωρίζουν τη μακροπρόθεσμα, μέσο πρόθεσμα, θα εξοικονομήσουν χρήματα, δεν έχουν το αρχικό κεφάλαιο, δεν έχουν οικονομίες και δεν έχουν δυνατό, μεγάλη επιστοληπτική ε, ικανότητα για να μπορέσουν να συλλέξουν το κεφάλαιο. Είναι πρόβλημα των ανθρώπων με χαμηλό Τρίτο πρόβλημα. Έχουμε και το δίλημα ποιο πληρώνει για, το, για την επένδυση για ενεργειακή απόδοση. Ο σπιτρονικοκύρης ή ο νοικιαστής. Αν ωφελείται ο ένας και όχι ο άλλος. Λέει ο νοικοκύρης πληρώνω για την ανακαίνιση, ε, μόνωση κλπ. Αλλά δεν μου επιτρέπεται να αυξήσω το νίκη. Και ο ένικος μπορεί να πει γιατί να κάνω εγώ κάτι, γιατί αυτό ωφελεί μόνο τον σπιτονικοκύρη που αυξάνει την αξία του ακινήτου του. Τώρα, οι πολιτικέ για την ενεργική αποδοτικότητα. Είπαμε για του στα εμπόδια πριν. Λοιπόν, τι πολιτικέ υπάρχουν ξεπεράσουμε τα εμπόδια. Έχουμε τρει ομάδε πολιτικών. Γενικέ πολιτικέ για ενεργική αποδοτικότητα συγκεκριμένες πολιτικές που απευθύνονται στα φτωχά νοικοκυριά και κοινωνικές πολιτικές που περιγράφονται άριστα και περιγράφει κανένα από τον συνάδελφο εδώ, τον Βενιαμίν Γκρενιέ. Οι κοινωνικές πολιτικές ανακουφίζουν γρήγορα τα προβλήματα, τον κίνδυνο της ενεργειακής ένδυας, γιατί πληρώνει το λογαριασμό. Οι γενικές πολιτικές. Και αυτές αντιμετωπίζουν το γενικό πρόβλημα της ενεργικής αποδοτικότητας. Δυστυχώς όμως δεν φτάνουν το κομμάτι αυτό του πληθυσμού που έχει πολύ χαμηλό εισόδημα. Και μόνο οι ειδικέ πολιτικές που απευθύνονται προς αυτοχάνικα κυριά είναι αυτές οι πολιτικές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Να οδηγήσουν σε κοινωνικά ωφέλη. Ε, δυστυχώς υπάρχουν ελάχιστες τέτοιες πολιτικές στην Ευρώπη. Ελάχιστες χώρες εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές. Οι άλλες χώρες δεν τις εφαρμόζουν. Κάποιες εκτιμήσεις βλέπετε εδώ. 50 με 120 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από ενεργειακή ένδυα στην Ευρώπη. 25 με 55 εκατομμύρια νοικοκυριά αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό. Και τα επιτυχή προγράμματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος έχουν επενδύσει κατά μέσο όρο από 2.500 μέχρι 5.000 ευρώ ανά νοικοκυριό για να βοηθήσουν τη βελτίωση της ενεργικής αποδικότητας του κάθε σπιτιού. Τώρα, χοντρικά, δεν τρέχουμε μελέτη, κάποια εκτίμηση χοντρική είναι αυτή. Κάναμε εκτίμηση συγκρίνοντας στοιχεία που έχουμε. Τάξη μεγέθους. 55 με 110 ε, ε, εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις για να λύσουμε το πρόβλημα της ενεργειακής ε, αποδοτικότητας στην οικοκαιριά. Εν γέννη. Αν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης. Πάμε τώρα στις συστάσεις για την, τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν. Εστιαστήκαμε επί έξι γενικών συστάσεων. Και δίνουμε και κάποιες λεπτομέρειες. Πρώτον, πρώτη σύσταση. Είπε η δόκτωρ Πετρόβα ότι η συζήτηση για την ενεργειακή ένδυα άρχισε σχετικά πρόσφατα, πριν από κάποιες δεκαετίες, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και ευτυχώς έχει διαδοθεί το θέμα σε όλη την Ευρώπη. Και συζητούμε το θέμα της ενεργειακής ένδυας. Όμως δεν υπάρχει κοινός ορισμός της ενεργειακής ενδίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσης και κοινό ορισμός των ευαλώτων καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν υπέρ και κατά. Ποιο είναι το συμπέρασμά μας. Καλύτερος είναι ένας κοινό ορισμός καλύπτοντας ιδιαίτερα τις διαφορές που ισχύουν στα διάφορα κράτη και γεωγραφικές περιοχές. Εκεί τα κράτη-μέλη μπορούν να καθορίσουν καλύτερα την ενεργειακή ένδυα όσον αφορά τι ιδιαιτερότητε των χωρών. Χρειάζεται όμω και κοινό ορισμό. Γιατί χρειάζεται κοινό ορισμό. Μόνο αν έχουμε κοινό ορισμό, νομικό κοινό ορισμό, μόνο τότε οι ευρωπαϊκέ οδηγίε μπορούν να είναι ακριβεί ε, του τι δέον γενέστε για την ε, επίλυση του προβλήματο. Η οδηγία για την αποδοτικότητα που αναδιατυπώνεται τώρα και η οδηγία την ενεργειακή επίδοση των κτηρίων Αυτές οι οδηγίες θα οδηγήσουν επίσης στη νέα, στο νέο ορισμό. Δεύτερος, ε, δεύτερη σύσταση. Έχουμε κοινωνικά ωφέλη, τα συζητήσαμε. Πέραν αυτό, πρέπει να λύσουμε και ένα πρόβλημα άλλο. Τη ενεργειακή αποδοτικότητα στα φτωχά νοικοκυριά, αν θέλουμε να πετύχουμε του στόχου μα για το κλίμα, για το 2030 και το 2050. Ποιο είναι το θέμα. 36% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακο προέρχονται από τον τομέα των νοικιακών, τη της αν θέλετε, από τα σπίτια. Αν θέλουμε να φτάσουμε, να πετύχουμε του στόχους για το κλίμα, όλα τα νοικοκυριά, φτωχά, με χαμηλό εισόδημα, πλούσια νοικοκυριά, όλα τα νοικοκυριά, όλα τα σπίτια πρέπει να έχουν ενεργειακή αποδοτικότητα στο μέλλον. Τι σημαίνει αυτό, ότι τα φτωχά νοικοκυριά θα πρέπει και αυτά να έχουν ενεργειακή αποδοτικότητα. Άρα Δημιουργείται ανάγκη επιλύσεως του προβλήματος από διαφορετική γωνία, όχι μόνο από την ε, κοινωνική, αλλά μέσω ενεργειακής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τι συστήνουμε λοιπόν. Πρώτον, οι οδηγίες αναδιατυπώνονται για την ενεργειακή αποδοτικότητα και ενεργειακή επίδοση των κτηρίων. Θα πρέπει να υπάρχει τακτική υποβολή αναφορών από τα κράτη-μέλη και να καλύπτεται όλη η στέγαση να καλύπτω τόσο ιδιαίτερω τα φτωχά νοικοκυριά και τα προβλήματα που υπάρχουν, τα, οι φραγμοί που υπάρχουν σε κάθε χώρα για την επίτευξη ενεργειακή αποδοτικότητα στα φτωχά Η οδηγία ενεργειακή αποδοτικότητα απαιτεί από τα κράτη-μέλη ή θα έπρεπε να απαιτεί να, έχει, να έχουν υπό για ευάλωτε ομάδε ενεργειακή αποδοτικότητα, όπω τα φτωχά Μετά, η, η οδηγία για την ενεργειακή επίδοση των κτηρίων θα θέτει ε, κάποια όρια για τις ελάχιστες ενεργειακές επιδόσεις. Μετά, άλλη σύσταση. Ο σχεδιασμός των πολιτικών για ενεργειακή αποδοτικότητα. Θα πρέπει ε, ρητά να αναφέρει τα κοινωνικά ωφέλη. Όταν σχεδιάζουμε τις ενεργειακές πολιτικές για τα φτωχά νοικοκυριά ή εν γέννη, θα πρέπει ρητά να αναφέρουμε ότι αυτό οδηγεί σε κοινωνικά ωφέλη επίσης. Όχι μόνο ωφέλη για το κλίμα ο σχεδιασμός θα πρέπει να περιορίζει αντιπαραγωγικά αποτελέσματα. Δηλαδή, όταν καταναλώνεις λιγότερη ενέργεια, μειώνει το λογαριασμό σου, καταναλώνεις ενέργεια για άλλους λόγους. Αυτό είναι μια αρνητική συνέπεια, ίσως για κάποια νοικοκυρία αυτό δεν είναι κακό. Ανεβαίνει το βιωτικό επίπεδο. Ποια είναι η συγκεκριμένη σύσταση. Ότι οδηγεί η ενεργειακή αποδοτικότητα και για την η οδηγία ενεργειακή επίδοση των κτηρίων και η οδηγία την αντικειτοθεσία απαιτεί από τα κάτι μέλη να λάβουν υπόψη τα πλεονεκτήματα για την ενεργειακή αποδοτικότητα στην ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση. Πρέπει να προβάλλονται τα ωφέλη και να υπάρχει ανταλλαγή των απόψεων και των ε, πορισμάτων περιθετικών αποτελεσμάτων μεταξύ κρατών μέλων. Να μαθαίνει μια χώρα την άλλη. Τέταρτον, τέταρτη σύσταση. Πλαίσιο πολιτική που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη μέτρα που καλύπτουν τους φραγμούς και τα προβλήματα που υπάρχουν για τα φτωχά νοικοκυριά, για τα ευάλωτα νοικοκυριά εν γέννη. Και τι συστήνουμε. Η οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα και η οδηγία για την ενεργειακή επίδοση των κτηρίων θα πρέπει στο προήμιο να φέρονται στα προβλήματα και εμπόδια και να απαιτεί το κράτη-μέλη αυτέ τι στοιχείε να τραβάνουν υπόψη στρατηγικέ για την ανακαίνιση κτηρίων, να έχουν όρια για, την, για, τους, ε, το μίστομα για κάποια κτίρια με χαμηλό επίπεδο ε, ενέργειας στην Ουτρέχτη, στην οργάνωση στέγασης, στην ΠΟΕΞ, εκεί έχουν ανακαινιστεί κτίρια με, που ε, εκτιστήκαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που είχαν πολύ χαμηλή και αποδοτικότητα. Έγινε ανακαίνιση χωρίς να ψηθεί το νίκη για τους ενοικιαστές και λειτουργήσε το σύστημα. Άρα, σωστή ενημέρωση χρειάζεται. Θα πρέπει τα ωφέλη να κοινοποιούνται σε όλου του εμπλεκομένου φορεί. Τελευταίε δύο συστάσει. Και ίσω σημαντικότερε. Η επιλογή συγκεκριμένων πολιτικών είναι καλύτερο να αφαιθεί στα χέρια των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει πρώτα απ' όλα να εφαρμόσουν διαθετικά προγράμματα, δομικά προγράμματα και πολιτικέ. Όχι απλώ μικρά προγράμματα, διαθετικέ πολιτικέ που υπάρχουν στι Ηνωμένε Πολιτείε και στη Νέα Ζηλανδία. Πολύ επιτυχή παραδείγματα. Στην Ευρώπη έχουμε πολύ καλά παραδείγματα. Έχει αναφερθεί ένα παράδειγμα από τον συνάδελφο, τον ήδη. Και η Τζούντι ανέφερε άλλο παράδειγμα. Για το παράδειγμα της Ιρλανδίας. Και πρόγραμμα για τη σκοτία υπάρχει και στη Γερμανία. Ήδη λοιπόν εμπεριέχονται εκεί στοιχεία που δείχνουν ότι μπορεί να πετύχει πολιτική για την ενεργειακή αποδοτικότητα των φτωχών οικοκυριών. Δίνονται σωστέ πληροφορίε στα φτωχά νοικοκυριά. Μετά έλεγχη για το ενεργειακό θέμα. Δωρεάν έλεγχη. Για να καθορίζεται τι μπορεί να βελτιωθεί σε ένα σπίτι. Τρίτον, βοήθεια στην ανακαίνιση να δίνονται χρήματα. Είτε δωρεάν χρηματοδότηση, είτε μερική χρηματοδότηση. Αλλά κάποια οικονομική ενίσχυση να δίνεται για να γίνει η ανακαίνιση. Θα πρέπει να ξεκινάμε από τη μόνωση στα σπίτια. Όχι με την αντικατάσταση ψυγείων, Φερρυπίν. Διότι αν αντικαθιστούμε συσκευές, και συσκευές, δεν πετυχαίνουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα. Τέλος τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τα διαθετικά μία κάποια, κάποιους πόρους από άλλα ταμεία της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Από αυτά τα ταμεία να παίρνουν χρήματα και να χρησιμοποιούν τα χρήματα για τη χρηματοδότηση των προαναφερθέντων μέτρων. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο και εγώ πρέπει να πω ότι πολύ καλή αυτή η ομιλία και παρουσίαση και τώρα μπορούμε να περάσουμε στην συζήτηση ανταλλαγή ερωτημάτων και απαντημάτων. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ζητήσω από τους συντονιστές ή τους αντικαταστάτες τους. Πολλοί βέβαια δεν είναι παρόντες, αλλά καταρχή η κυρία Γκρίφιθ από τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Ευχαριστώ Γιαζή και ευχαριστώ αυτούς που έκαναν τις παρουσιάσεις. Ουσιαστικά κάνετε κήρυγμα σε αυτούς που ήδη είναι πιστοί σε σχέση με τα θέματα αυτά. Εμείς είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα στην έκθεσή μας για την προστασία των καταναλωτών που αναφέρεται στο θέμα αυτό. Εμείς ως σοσιαλιστές και κάποιοι από τους συναδέλφους μου είναι εδώ που έχουν συμμετάσει. εμείς έχουμε αναπτύξει ήδη μια πολιτική για την ενεργειακή ένδυα εγώ έρχομαι από τον Αγγλικό Βορρά, από την περιοχή του Λίβερπουλ, όπου πολλοί πολίτες πρέπει να διαλέξουν μεταξύ του να αγοράσουν φαΐ και του να θερμανθούν. Στη χώρα μας έχουμε αυτό το πρόβλημα, ενώ αντίθετα μου είπε ένας, Ιταλός, ένας Ισπανός συνάδελφος, πεθαίνουν άνθρωποι το καλοκαίρι γιατί δεν έχουν το, την, ε, τα λεφτά να χρηματίσουν κλιματιστικά. Επομένως αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε και το αναφέρετε κι εσείς είναι να τονίσουμε ότι η ενέργεια δεν είναι ένα αγαθό <clears throat> και μόνο. Πρέπει να είναι ένα βασικό ανθρώπινο κοινωνικό δικαίωμα. Δεν έχουμε επιτύχει ακόμα να συνειδητοποιήσουμε όλο τον κόσμο για το θέμα αυτό, αλλά συνεχίζουμε τις προσπάθειε μα γιατί οι συστάσεις σας δίνουν το σωστό πλαίσιο για όλη την νομοθεσία. Αν θεωρηθεί βασικό κοινωνικό δικαίωμα η ενέργεια, πολλά προβλήματα θα αλλάξουν. Η προσπάθειά μας είναι λοιπόν να πείσουμε τους καταναλώτες να ξέρουν ποια είναι η φθηνότερη πηγή ενέργειας. Δεν έχουμε πετύχει ακόμα και αυτό το μέτρο, αλλά προσπαθούμε ακόμα. <clears throat> Ξέρουμε ότι μία αύξηση κατά 1% σε ενεργειακή ε, απόδοση μπορούν να οδηγήσουν σε 3 εκατομμύρια σπίτια τα οποία μπορούν να ανακαινιστούν και οι κάτοικοι τους να βγουν από την ενεργειακή από, την ενεργειακή ένδια. Πολλέ φορέ οι πιο φτωχοί είναι αυτοί που ζουν στα σπίτια με περισσότερα ρεύματα και χειρότερη ε, ενεργειακή μόνωση. Και είπατε επίση και για το θέμα των ιδιοκτητών των σπιτιών που νοικιάζονται Πώς μπορούμε να τους δώσουμε κίνητρα ώστε να μην πρέπει να πληρώσει ο Νικάρης. <clears throat> Πώς μπορούμε λοιπόν <clears throat> να κινητοποιήσουμε και τους τοπικούς παίκτες στο θέμα αυτό. Η COP21 στο, Μαρακέ, στο Μαρακές. Σας λέω και πάλι δεν είναι ένα θέμα μονάχα κοινωνικών λύσεων, είναι αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της σωστής κοινωνικής πολιτικής. Ξέρετε ότι η Κομισιόν έχει αποφασίσει να έχει ένα κατά κάποιο τρόπο ισολογισμό ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως απαιτεί ένα κοινό για την ενεργειακή ένδυα, <clears throat> καλή συνεχή ε, δεδομένων. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο αυτό. Πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε τη μεταλαμπάδευση βελτίστων πρακτικών αν ξέρουμε ότι οι πρακτικέ αυτέ τη Σκωτία και της Ουτρέχτη και τη Γερμανία μπορούν να είναι οι καλύτερε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι και η Βουλγαρία χρησιμοποιεί αυτέ τι πρακτικέ και το Λίβερπουλ το χρησιμοποιεί. Έτσι με τον τρόπο αυτό μπορούμε όταν έχουμε λύσεις οι οποίες είναι σωστές και οικονομικά να χρησιμοποιούνται από όλους <clears throat> ώστε να υπάρχει συνειδητοποίηση αυτών των λύσεων. Το ξέρω γιατί εγώ εκπροσωπώ γυναίκες που νιώθουν παρικό όταν βλέπουν το λογαριασμό του ηλεκτρικού του στο σπίτι τους και πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν άνθρωποι ευάλωτοι που να τους κόβουν το ρεύμα. Ευχαριστώ, Τέρεσα, λοιπόν. Από το ECR, ο κ. Χένκελ, ο αντιπρόεδρος μας. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι πιστοί όλοι αυτοί που άκουσαν τη συνταχέ σας. Έχω κάποιο πρόβλημα με την δική σας προσέγγιση, λέει ο κ. Χέγκελ. Νομίζω καταρχήν, <clears throat> νομίζω ότι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι αυξάνουν τις ενεργειακές τιμέ είναι αυτοί οι οποίοι τώρα ανησυχούν για το αποτέλεσμα που έχουν αυτέ τις τιμέ στου φτωχότερου. θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι υπάρχει μια τέτοια σύνδεση. Δεν άκουσα κάτι τέτοιο να λέγεται από τους ομιλητές μας. Πιστεύω επίσης ότι είναι ατυχές το ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην ενέργεια, αλλά είναι εξίσου σημαντικό και αρνητικό το ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να αγοράσουν φαΐ ή ρούχα ή δεν μπορούν να στεγαστούν. Έχουμε τώρα <clears throat> σχέδια αντιμετώπισης της φτώχειας για όλα αυτά τα στοιχεία. Αλλά πρέπει να είναι χωριστά αυτά. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια κοινωνική πολιτική αντιμετώπιση ένδυα, αυτό είναι σωστό. Χρειαζόμαστε μια πολιτική περιβάλλοντος για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε ενεργειακές πολιτικές, αλλά αν τώρα αρχίσουμε να αναμειγνύουμε την κοινωνική πολιτική, πολιτική καταπολέμησης της ένδειας με την ενεργειακή πολιτική, θα οδηγηθούμε σε πάρα πολύ δραστική και υπερτροφική κρατική παρέμβαση. <clears throat> Δεν είμαι πεπισμένος λοιπόν ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Αυτό ευχαριστώ πολύ λέει και ο πρόεδρος. Ο Κλοντ Τσούρμες έχει το λόγο από τις πρόασους. Ευχαριστώ Γερζή. Το πρώτο μήνυμά μου είναι ότι η ένδια είναι ένδια. Έχουμε λοιπόν προβλήματα στην Ευρώπη με την ε, λανθασμένη αντιμετώπιση της κρίσης των, της Lehman Brothers στις ΗΠΑ, μια κρίση η οποία έριξε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν φτωχοί σε μια κρίση ένδυας. Ας δούμε λοιπόν το ευρύτερο πλαίσιο. Έχουμε επίσης το ειδικό θέμα της ενεργειακής ένδυας <clears throat> που εκεί βλέπω δύο υποπεριοχές. Πρώτα απ' όλα η ειδική κατάσταση των χωρών που ήταν στο παρελθόν της Σοβιετικής Ένωσης που είχαν μια κουλτούρα αναποτελεσματικότητας με μια κουλτούρα τεχνητά επιδοτούμενων χαμηλών τιμημάτων ενέργειας <clears throat> και που σήμερα δεν έχουν φτάσει φυσικά την αγοραστική δύναμη της Γερμανίας ή της Δανίας. Γι' αυτό αυτό το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε είναι να προχωρήσουμε κυρίως σε ένα κοινό ορισμό αλλά να εξασφαλίσουμε να μην ακολουθήσουμε και την αγγλική ε, <clears throat> προσέγγιση ότι όλοι μπορεί να είναι ενεργειακά φτωχοί ανεξάρτητα από το που βρίσκονται. Πρέπει να χαράξουμε και μια πολιτική ενεργειακής απόδοσης στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή αυτή η πολιτική αφορά τα νοικοκυριά της, ε, των υψηλότερων τάξεων που έχουν χρήματα στην τσέπη τους και πρόσβαση στο ίντερνετ. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ αυτά που είπε ο Σέρχιο για το πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση στο κεφάλαιο και πώς μπορούμε να έχουμε πληροφορίες οι οποίες θα είναι εύκολα προσβάσιμα, προσβάσιμοι από ανθρώπους που δεν έχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα και που είναι διαφορετική από τις φόρμες που έχει το πρόγραμμα για την ενεργειακή απόδοση. Θέλουμε μια πιο ευφυή Ευρώπη σε επίπεδο ενεργειακής απόδοσης και θα πρέπει να φέρουμε τα καλύτερα μυαλά στην Ευρώπη από κοινού για να, για να μας πούν πώ θα αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή ένδυα και χρειάζεται και καλύτερη χρήση του ευρωπαϊκού προπολογισμού, του, των διαφορετικών ταμείων, του Ταμείου Γιούγκερ, του Κοινωνικού Ταμείου στην Ανατολική Ευρώπη, γιατί η Ανατολική Ευρώπη, για του ιστορικούς λόγους που ανέφερα προηγουμένω έχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε για να προλάβει την υπόλοιπη Ευρώπη. <clears throat> πρέπει λοιπόν να δώσουμε περισσότερα διαφορετικά ταμεία, περισσότερη χρηματοδότηση από το ΕΦΣΥ και περισσότερα κονδύλια από το Κοινωνικό Ταμείο, ώστε η Ανατολική Ευρώπη να μπορέσει να ανανεώσει ενεργειακά τα κτίρια της, ιδίως με το να μπορούν να έχουν πρόσβαση κεφάλαιο για την ενεργειακή αναβάθμιση. Χαίρομαι που χθε η Κομισιόν ανέφερε ένα νέο σχέδιο εργασία για την οικολογική σχεδίαση. Το να έχουμε αποτελεσματικέ ενεργειακέ συσκευέ είναι ο καλύτερο τρόπο να μπορέσουμε να μιλήσουμε το τίμημα τη ενέργεια, το κόστο τη ενέργεια και χαίρομαι που ο κύριο Τίμερμαν έχει αναγνωρίσει ότι το θέμα της οικολογική σχεδίαση και τα συναφή μέτρα μπορούν να παίξουν μεγάλο ρόλο και να προωθήσουμε λοιπόν οικολογικές συσκευές, οι ηλεκτρικούς μηχανισμούς κτλ. Ο κύριος Σιδικιώτης από την ΚΟΕ. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, νομίζω είναι ευχαριστήσω τους συζητητές. Ε, είναι σωστή η διαπίστωση ότι ε, μεγάλα τίμηματα του πληθυσμού ε, έχουν διορισμένη στην ενεργειακή ένδυα ε, δεν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να καλύψουν τις ε, ενεργειακές τους ανάγκες είτε αυτό αφορά ηλεκτρισμό ή θέρμαση εγώ θα έλεγα επειδή προέρχομαι από τον Νότο σε μερικές περιπτώσεις χρειάζεται σε εμά ε, ο κλιματισμός ε, το στο πρέπει να δώσουμε ένα ορισμό και συμφωνώ με τη συνάδελφο του, από το S&D τι είναι σήμερα ενέργεια είναι δημόσιο ανθρώπινο αναγκό είναι μια καθημερινή ανάγκη Άρα για να μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης για όλους σε φθηνή ενέργεια, δηλαδή επάρκεια σε ενέργεια και φθηνή. Είναι γι' αυτό που θεωρώ ότι τα μέτρα που έχετε αναφέρει δεν τα υποτιμώ. Κοινωνική πολιτική στήριξη δηλαδή των ευάλωτων ομάδων ή ε, ε χτίρια με ενεργειακή απόδοση. Δεν απαντούν όμως το κύριο. Κατά τη δική μας την άποψη όσο τα δίχτυα διανομής και παραγωγής της ενέργειας βρίσκονται σε ιδιωτικά χέρια, δεν θα αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια. Είναι για αυτό που εκείνο που χρειάζεται πάνω απ' όλα είναι τα δίχτυα και υποδομέ ε, να είναι δημόσια για να μπορούν να λαμβάνουν και το δημόσιο και το κράτος την ευθύνη του ε, ε απέναντι ε, στις πολίτες. Γιατί από τη στιγμή που σήμερα με τι οικονομικέ πολιτικέ που εφαρμόζονται, τι νεοφιλεύθερε πολιτικέ, τι πολιτικέ τη λιτότητα, όταν ο άνθρωπο δεν μπορεί να καλύψει τι βασικέ του ανάγκε ε, ε, ε, για να μπορεί να έχει καθημερινά φαΐ ή ακόμα και στέγαση, αντιλαμβάνεστε δεν θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει και τις ανάγκες στην ενέργεια. Πέραν από αυτό υπάρχουν και μέτρα που δεν φτάνει να δώσει στον άλλο μια, να του δίνει κάθε ε, ε, τόσο βοήθεια υπό την ανάγκη ότι το κράτο ασκεί κοινωνική πολιτική και δεν την υποτιμώ για να αντιμετωπίσει κάποιε ανάγκε. Εκείνο που χρειάζεται ο κόσμο είναι βοήθεια για να μπορεί ο ίδιο να έχει πρόσβαση ε, σε ευθυνή ενέργεια. Θα φέρω δύο παραδείγματα απλά από τι χώρε του Νότου. Στην Ελλάδα ε, σήμερα γίνονται, υπάρχουν περιοχές ε, πολλοί λόγω της κρίσης που είναι φτωχές. Υπάρχει δίχτυα φυσικού αερίου, όμως πολλά νοικοκυριά δεν έχουν τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν τον εξοπλισμό για να έχουν αυτή την πρόσβαση. Ε, άρα είναι κύριο να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν τον εξοπλισμό, όχι να λέμε ότι τα δίχτυα φτάνουν παντού. το δεύτερο παράδειγμα που θέλω να φέρω είναι κάτι που έχουμε εφαρμόσει στην Κύπρο. Είναι το σύστημα του, ένα σύστημα net metering που λέγεται συμψηφισμό. Δηλαδή, βοηθούμε νοικοκυριά που δεν έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να εγκαταστήσουν συστήματα φωτοβολταϊκό στα σπίτια τους να δίνουν και να συνδεδεμένα με τα δίχτυα και μέσα από την ε, παραγωγή ενέργειας και τον συμψηφισμό να πληρώνουν πάρα πολύ ελάχιστο ποσό για την ηλεκτρική ενέργεια, γιατί γίνεται ένας συμψηφισμός. Άρα το συζητούμενο είναι να ε, βοηθήσουμε τα νοικοκυριά για να εγκαταστήσουν ε, τέτοιους ε, υποδομές για να μπορούν να έχουν πρόσβαση. Και το τελευταίο, από, το τελευταίο που θέλω να πω είναι οι ενεργειακές νησίδες. Υπάρχουν κράτη-μέλη, υπάρχουν περιοχές στην Ένωση που δεν είναι συνδεδεμένες με τα μεγάλα δίχτυα ενεργειακά. Άρα δεν μπορούν να έχουν φθηνή ενέργεια. Να φέρω δύο παραδείγματα. Είναι Κύπρος και Μάρτα που είναι νησιά, αλλά υπάρχουν και άλλες ορεινές περιοχές και νησίδες ε, που είναι αναγκασμένες να εισάγουν μόνο συμβατικά καύσιμα και με αποτέλεσμα η ενέργεια να είναι σε ψηλέ τιμέ. Διότι δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση ε, στα ευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα και είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη ε, και όχι μόνο τα κράτη-μέλη. Ε, από μόνα του. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κόλιτσεκ, αντιπρόεδρος. Κόλιτσεκ. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος από τους Πράσινους που τώρα μιλάει με τον ε, πρόεδρο ο εκπρόσωπος των Πρασίνων, νομίζω ότι έχει δίκιο. Είπε ότι στις ανατολικές χώρες υπήρχε φτηνή ενέργεια. Μα ακριβώ παντού πρέπει να είναι φτηνή ενέργεια και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στο Βέλγιο. Ακόμα και στην Αγγλία ήταν φτηνή η ενέργεια γιατί είχαν τους δικούς τους ενεργειακούς πόρους. Αν λοιπόν συγκρίνουμε τις δυνατότητες του κόσμου, πρέπει να δούμε το μέσο όρο των μισθών. Στην Τσεχία ή στη Βουλγαρία, μόνο το 1 τρίτο του κόσμου έχει το μέσο όρο των εισοδημάτων. Οι άλλοι έχουν χαμηλότερο. Αν συγκρίνουμε τους μισθούς της Βουλγαρίας και της Τσεχίας με τους μισθούς της δυτικές χώρες, τότε Πράγματι, οι περισσότεροι άνθρωποι στις ανατολικές χώρες δεν είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε νέες τεχνικές. Από την άλλη μεριά, το πρόβλημα με το καύσωνα ε, δεν είναι μόνο στο Νότο. Στο Λίβερπουλ, για παράδειγμα, ήμουνα και υποφέραμε. Τα κτίρια λοιπόν πρέπει να έχουν καλύτερη μόνωση, καλύτερα παράθυρα, αλλά το κύριο πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει, για την ενεργειακή ένδυα είναι η μισθή. Αν συγκρίνουμε τους μισθούς, διοπιστώνουμε ότι υπάρχουν διαφορές 1 προς 10 και είναι αυτό ένα χάσμα το οποίο αυξάνει. Πρέπει να περιμένουμε λοιπόν να μικρύνει το χάσμα αυτό και μόνο τότε μπορούμε να μιλήσουμε για ένα κοινό ορισμό της ενεργειακής ένδυας. Γιατί δεν μπορεί κανείς να συγκρίνει πλούσιες με φτωχές χώρες. Στην Βουλγαρία 50% του κόσμου είναι ενεργειακά φτωχός, ενώ στη Γαλλία, στις χώρες Μπενελούξ και αλλού, όπου η μισθή είναι πολύ πιο ψηλή, Εκεί βλέπουμε ότι τα μέτρα μόνωση στα διπλά τζάμια κλπ. λειτουργούν. Ή τα φωτοβολταϊκά, όλα αυτά τα μέτρα είναι εφικτά στις δυτικές χώρες, γιατί ο κόσμος έχει χρήματα να τα πληρώσει. Η κυρία Σπυράκη, κύριε Σπυράκη, λυπάμαι Μαρία, λυπάμαι, γιατί δεν σας βρήκα νωρίτερα έξω. Η κυρία Σπυράκη. Δεν πειράζει, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ όλους τους συμμετέχοντες εδώ στην παρουσίαση αυτή, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ γρήγορα. Και δεύτερον, το θέμα για μένα είναι πόσο γρήγορα μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα πρέπει να ανταλλάξουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Πράγματι, πρέπει να συνεχίσουμε να ανταλλάσσουμε μεταξύ μας τις βέλτιστες πρακτικές, να συζητάμε για καλύτερα κτίρια, καλύτερη στέγαση. Και προς αυτό το σκοπό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε βέβαια και κονδύλια από τα ταμεία, αλλά και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Είναι ενδιαφέρον το... η εμπειρία των Παρισίων με 60.000 διαμέρισματα. Πρέπει να δούμε πώς τα κατάφεραν εκεί στη Γαλλία. Και έπειτα, το κόστος της ενέργειας και ενεργειακή μας αγορά. Για το θέμα της Ελλάδας, η ιδιωτικοποίηση της εταιρείας ηλεκτρισμού είναι ένα ζήτημα που πρέπει να παρακολουθήσουμε στενά και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί υπάρχουν ενστάσεις ακόμα και από υπουργού μέσα στην κυβέρνηση. Άρα λοιπόν πρέπει να βλέπουμε και την ομοθεσία, αλλά και τα συνέπειε αυτής. Πρόεδρος, ευχαριστούμε Μαρία. Ωραία, εδώ τέλειωσαν οι ερωτήσεις. Οπότε σας παρακαλώ τώρα να απαντήσετε κάπως σύντομα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κυρία μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας και για τις ερωτήσεις σας. Θα ήθελα να πάω λίγο πίσω σε κάποια από αυτά που σας είπα πριν. Το πρώτο είναι ότι η ενεργειακή ένδια ίσως να μην έπρεπε να ονομάζεται έτσι. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το εισόδημα, και γι' αυτό μιλάμε για φτώχεια, έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες οι οποίοι συγκεντρώνονται και οδηγούν σε μία έλλειψη υλικών αγαθών. Όταν μιλάμε για την ε, φτώχεια στα τρόφιμα, μιλάμε για τρόφιμα, αν μπορούν ή δεν μπορούν να αγοράσουν ε, τρόφιμα οι άνθρωποι. Όταν όμως μιλάμε για την ενεργειακή ένδυα, δεν μιλάμε μόνο για το εισόδημα, μιλάμε και για το σπίτι σου. Μιλάμε για το αν είσαι σε θέση να έχει μια κανονική ζωή μέσα σε μια κοινωνία. Συνεπώ, και το βλέπουμε παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό, και όχι μόνο στην Ανατολική ή στην Νότια Ευρώπη, ότι ο κόσμος με μεσαία εισοδήματα, αν παγιδευτεί σε μια αγορά, για παράδειγμα, ενοικίασης, τότε μπορεί να διαπιστώσουμε ότι δεν μπορεί να βοηθηθεί και γι' αυτό στερείται διάφορα αγαθά. Και ακόμα και αν έχουν πιο υψηλά εισοδήματα, τελικά δεν θα φτάνουν για να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους. Το δεύτερο που θέλω να αναφέρω είναι τα νοικοκυριά χαμηλών εισοδημάτων. Βεβαίω η έρευνα δείχνει ότι στις ηθικές κοινωνίες πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα νοικοκυριά αυτά και όχι μόνο γιατί πρέπει και αυτά να έχουν μια φυσιολογική ζωή σε κανονικά σπίτια, αλλά γιατί και τα ωφέλη της ενεργειακής ε, απόδοσης είναι πολλαπλά, όπως είπε και ο συνάδελφος. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, λοιπόν το ωφέλη στην υγεία. Η ακαδημαϊκή έρευνα έχει δείξει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε κοινωνικές κατοικίες μερικές φορές δεν πρόκειται μόνο για εξοικονόμηση άνθρακα. Δεν χρησιμοποιούν οι άνθρωποι αυτοί τόση πολύ ενέργεια. Δεν μπορούν να επιτρέψουν σε αυτούς τους να καταναλώνουν πολύ ενέργεια. Αν όμως βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των σπιτιών τους τότε θα κερδίσουν και τα δημόσια συστήματα υγείας, γιατί θα μειωθεί το κόστος για την υγεία. Οπότε όταν μιλάμε για την ενεργειακή ένδια, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα ωφέλη σε διάφορους ε, τομείς, αν αντιμετωπιστεί αυτή δηλαδή. Τώρα για τις θέσεις σοσιαλιστικές χώρες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Πρέπει να πω ότι πρέπει να αναγνωρίσω κάποιες από τις προσπάθειες που έγιναν σε κάποιες από αυτές τις χώρες για την ενεργειακή απόδοση κυρίως. Και πραγματικά θέλω να αναφέρω την ιδέα της Έλενα Σούσπορνα στην Τσεχία, όπου η χώρα έδωσε χρηματοδότηση για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων. Ένα πρόβλημα πάντως είναι ότι οι αποφάσεις που λήφθησαν στην περίοδο μετά τον σοσιαλισμό είναι που επηρέασε τα πράγματα. Σε πολλές περιπτώσεις η στέγαση είναι παγιδευμένη σε ενεργειακά συστήματα τα οποία δεν είναι αποτελεσματικά. Είτε είναι περιφερειακά, είτε πρόκειται για τερικές σχέσεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, οπότε νοικοκυριά δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να χρησιμοποιήσουν την θέρμανση που δίνεται στη συγκεκριμένη περιοχή και το κόστος μερικές φορές είναι πολύ μεγάλο. Δεν έχουν την επιλογή δηλαδή. Σίγουρα πολλά έχουν ήδη γίνει, αλλά υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Κάτι άλλο ήθελα να πω. Για να πάω πάλι πίσω στην παρουσίασή μου στους έξι παράγοντες, ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι η ευελιξία του ενεργειακού συστήματος. Αν πάμε πίσω στον ορισμό, Κάποιος είπε ότι αν ακολουθούμε το 10% ε, μπορεί και η βασίλισσα της Αγγλίας να αποδειχτεί ότι είναι ενεργειακά φτωχή. Γιατί μπορεί να χρειάζεται πάνω από 10%. Αλλά εδώ επανέρχομαι στο θέμα της επιλογής. Πρέπει να έχουμε την επιλογή. Για κάποια νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γεγονός αυτό. Αλλά σε άλλες χώρες μέλη δεν μπορούν τα νοικοκυριά να αλλάξουν από ένα ενεργειακό σύστημα και να πάνε σε ένα άλλο. Στηρίζω λοιπόν την ιδέα αυτή και νομίζω ότι είναι η σωστή στιγμή για να μιλήσουμε για την ενεργειακή ένδυα, κυρίως αν λάβουμε υπόψη μας τις αλλαγές που γίνονται στην ενέργεια με τις διαδικασίες έλλειψης και μείωσης της κατανάλωσης του άνθρακα. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. επόμενο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κι εγώ. Θέλω να επανέλθω σε κάποια σημεία που ακούσαμε στη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, και εγώ πιστεύω ότι η ενεργειακή ένδια ω έννοια είναι χρήσιμη. Γιατί μιλάμε για αποδοτικές πολιτικές ενεργειακή απόδοση, μιλάμε για κοινωνικές πολιτικές και μπορούμε αυτά να τα κρατήσουμε χωριστά αν θέλουμε, αλλά εγώ νομίζω ότι κάπου αυτά τα δύο συνδέονται και είναι ακριβώ την ενεργειακή ένδια. Προσπαθούμε να κάνουμε πιο αποδοτικά τα, ε, ενεργειακά τα κτίρια, αλλά αυτό απαιτεί πάρα πολλά χρήματα. Οπότε το θέμα είναι πώς καθορίζουμε προτεραιότητες. Και αν μιλάμε για ενεργειακή ένδυα, τότε θα βάλουμε σαν προτεραιότητα τα κονδύλια για την βελτίωση των κτηρίων, για να βοηθήσουμε και τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων που ζουν σε αυτά. Συνεπώς πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμη αυτή η έννοια. Έπειτα, όσον αφορά τις αιτίες της ενεργειακής ένδυας, κάποιοι είπαν στη συζήτηση ότι είναι οι αλλαγές που γίνονται, είναι η πράσινη ενέργεια, είναι η λιτότητα. Είναι όμως και θέματα ε, πολιτικών αποφάσεων. Οπότε, αν, ακόμη και να αφήσουμε απ' έξω τις πολιτικές, η Διεθνής ε, Υπηρεσία Ενέργειας έχει στην τελευταία της έκθεση, και τώρα που να είναι θα έρθει και μια νέα, λέει ότι αυξάνονται οι τιμές της ενέργειας. Ακόμα και αν έχουμε αποπληθωρισμό, παρόλα αυτά η τιμή της ενέργειας αυξάνει. Οπότε τα νοικοκυριά τα οποία είναι χαμηλών εισοδημάτων ή δεν κατοικούν σε κτίρια ενεργειακά αποδοτικά θα υποφέρουν ακόμα περισσότερο από την αύξηση των τιμών. Άρα γι' αυτό χρειάζεται βελτίωση των ε, πολιτικών μας όσον αφορά το κλίμα και οι κοινωνίες να γίνουν ε, περισσότερο αντοχής τώρα που αλλάζουμε και περνάμε από τα ορυκτά σε άλλες μορφές ενέργειας. Τώρα το είπε και η κυρία Πέτροβα Εντάξει, ναι, ανάλογα με το τι ορισμό χρησιμοποιούμε για την ενεργειακή ένδια, μπορούμε να καταλήξουμε ότι η Βασίλισσα της Αγγλίας είναι ενεργειακά φτωχή. Πάντως, στο Μπάκεχαμ θα έπρεπε να αναρωτηθούμε τι κόστος χρειάζεται η θέρμανσή του σε κάποιο επίπεδο. Αν έπρεπε να πληρώσει για την ε, για το κόστος αυτής της θέρμασης, πολύ πιθανό να μην μπορούσε η Βασίλισσα. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερη έρευνα για να έχουμε την ακρίβεια που χρειαζόμαστε στους ορισμούς κτλ. Και πάντα πρέπει να καταλήγουμε σε ένα συμβασμό. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γκράινερ, τώρα ο κύριος Σουγκάρντε. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα μία σκέψη μου. Όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα βιολογικά έχουν ε, την ανάγκη για δύο φορές περισσότερο από όσοι υπόλοιποι, γιατί έχουν ακριβώς χαμηλό εισόδημα. Οπότε τι κάνουμε. Αυξάνουμε την κοινωνική βοήθεια για τα άτομα αυτά ή διορθώνουμε τη βιολογική δυσλειτουργία που εμποδίζει τα άτομα αυτά να λειτουργήσουν κανονικά, γιατί υποφέρουν περισσότερο η υγεία τους και τέτοια. Οι διαφορές στους μισθούς εννοείται ότι παίζει επίσης ρόλο, γιατί τα άτομα αυτά έχουν χαμηλότερα εισοδήματα από τους άλλους, άδικο, αλλά πάντων δεν είναι αυτό που αναλύουμε τώρα. Απλώς σκεφτείτε αυτό το ειδικό πρόβλημα. Μικτές πολιτικές, δεν ξέρω, οι πολιτικοί πρέπει να το συζητήσουν αυτό, θα το κάνετε δίχως άλλο. Αλλά υπάρχουν και πιο θεμελιώδη ζητήματα που είναι η πηγή, οι αιτίε της ενεργειακής ένδυας που δεν είναι μόνο τα χαμηλά εισοδήματα. Έρχομαι στις ενεργειακές, ενεργειακές τιμές που είναι και αυτός πυλώνας και αιτία. Και υπόθηκε ότι είναι πολύ ψηλές οι τιμές. Ενεργειακές τιμές λοιπόν. Υπάρχει δυνατότητα τώρα με την ενεργειακή απόδοση να υπάρχει συνέπεια και επί των τιμών. Η μεταρρύθμιση στον ηλεκτρισμό γίνεται τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και στη μεταρρύθμιση αυτή για τον ηλεκτρισμό υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το πώς πρέπει να οργανωθεί ο κλάδος. Και τίθεται το θέμα της ευελιξίας. Τι κάνουμε λοιπόν για να δώσουμε περισσότερη ευελιξία στο σύστημα, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί και στην ζήτηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Υπάρχουν περισσότερες πηγές, να συνδυαστούν οι πηγές, να υπάρχει ευελιξία στον κλάδο. Τελικά όμως αυτό καταλήγει στο να έχουμε πιο ακριβή ενέργεια. Υπάρχουν όμως και άλλες ε, επιλογές στην ευελιξία. Δεν ξέρω αν θα επιλεχθούν, αλλά υπάρχουν. Ενεργειακή απόδοση είναι ένας παράγοντας. Διασύνδεση. Το είπε ο βουλευτής από την Ελλάδα, νομίζω. Επίσης υπάρχει το θέμα της πρόσβασης στις υποδομές. Καλύτερη διασύνδεση λοιπόν και ενεργειακή απόδοση είναι δύο πολύ καλές επιλογές ευελιξίας που θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στη μεταρρύθμιση για τον ηλεκτρισμό. Και γιατί. Γιατί η ενεργειακή επάρκεια είναι το μέτρο εκείνο το οποίο επηρεάζει περισσότερο τις τιμές. Και κάθε επίδραση στις τιμές έχει τεράστια επίδραση στα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα γιατί οι δαπάνε ενεργειακέ για τα νοικοκυριά αυτά χαμηλών εισοδημάτων αναλογικά είναι πολύ μεγαλύτερα. Τώρα για την πρόσβαση σε κεφάλαιο. Ναι, πώ να έχουμε πρόσβαση σε κεφάλαιο. Εγώ σα είπα ήδη τα κοινωνικά ταμεία, τα Ταμείο συνοχή για τι αντικέ επενδύσει, περιφερειακή ανάπτυξη και κοινωνικό ταμείο. Ναι, βεβαίω, αυτά τα ταμεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αλλά όχι μόνο αυτά. Νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Αλλά όχι μόνο αυτά. Υπάρχουν και ταμεία που έχουν φτιαχτεί υπέρ της υγείας ή της ασφάλειας. Αν λοιπόν χαμηλή ε, κατανάλωση ενέργειας δεν βοηθάει την υγεία, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το Ταμείο για την Υγεία για να συνδράμουμε στα θέματα της ε, ενέργειας γιατί θα μειωθεί ο λογαριασμός για την υγεία. Όταν θα έχει καλύτερη υγεία ο κάθε καταναλωτής. Άρα λοιπόν υπάρχει επίσης το ταμείο για τους ηλικιωμένους ή για την ανανέωση των κτηρίων. Έπειτα η πληροφόρηση κάποιος τόπο ότι δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση. Πάρα πολύ καλό παράδειγμα του προγράμματος Κάριτας στη Γερμανία. Νίκιασαν άνεργους με κάποια εκπαίδευση και τους κατάρτισαν στα θέματα της ενεργειακής επάρκειας για τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί μιλάνε την ίδια γλώσσα. Ξέρουν πώς να επικοινωνήσουν και πώς να ενημερώσουν τον κόσμο, δεν έρχονται από ψηλά και δεν έχουν ιδέα. Ξέρουν να τους πούνε τι πρέπει να κάνετε, αυτό το ψυγείο να το αλλάξετε ή το άλλο. Είναι η σωστή σωστη γλωσσα και άρα παίρνουν τη σωστή πληροφορία οι άνθρωποι. Πολλά λοιπόν θέματα κοινή λογική θα μπορούσαν ε, να εφαρμοστούν κάπως πιο δομημένα. Και είναι εφικτό. Γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Έξοχε ομιλίε και ακριβείς απαντήσεις. Και από τους τρεις σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Σάσκα Πέτροβα, κύριε Βενιαμίν Γκράινερ και κύριε Σέζιο Γουάρτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. And now Τώρα παρευθύ στο επόμενο σημείο. Έχουμε καθυστερήσει. Ευρωπαϊκά πρότυπα. Εφαρμογή του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας πω ότι η Ήτρε συμμετέχει βάσει το άρθρο 54. Η ΙΜΚΟ είναι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα όσον αφορά το ICT για την πληροφορική και την πολιτική καινοτομία. Σε αυτά εξαρτώνται από εμά. Η είναι ο κ. Χέγκελ. και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπατε, η δική μας Επιτροπή θα ετοιμάσει γνωμοδότηση για την τυποποίηση ε, διαφόρων στοιχείων όσον αφορά την πληροφορική, την τεχνολογία, 5G ε, επικοινωνίες, ε, υπολογισμοί στον έφος, στο ηλεκτρονικό έφος, στοιχεία κλπ. Κυβερνοασφάλεια και βάσει του άρθρου 55 εμείς έχουμε αποκλειστικές αρμοδιότητες για αυτά τα θέματα και έχουμε και μεικτή αρμοδιότητα, κοινή αρμοδιότητα με την ΙΜΚΟ. Η γνωμοδότηση της ΙΤΡΕ θα καλύψει και την τυποποίηση και την πρωτοβουλία για την τυποποίηση όσον αφορά τον ορίζοντα 2020 και την πολιτική για την καινοτομία και το κοινό κέντρο ερευνών. Το σχέδιο εκθέσεως θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους. Θα στείλουμε πρόσκληση την επόμενη εβδομάδα για την πρώτη συνεδρίαση των σκιωδών και μετά θα αρχίσουμε τις επαφές με τις ε, πολιτικές ομάδες Αυτές οι προδιαγραφές για τον τομέα της πληροφορικής έχουν σαν στόχο τη διαλειτουργικότητα που είναι και η πεμπτουσία της ψηφιακής οικονομίας και βάση για τη δημιουργία τεχνολογικών βάσεων που επιτρέπουν την καινοτομία. Εθελοντική, σφαιρική και διαφανής τυποποίηση και σχετικός μηχανισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να είναι επιτυχής προσέγγιση για να έχουμε κοινά πρότυπα στην εσωτερική αγορά. Όμως, θα πρέπει να δούμε ότι κάποια πρότυπα έχουν ήδη θεσπιστεί και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Όμως αυτά τα πρότυπα ξεπερνούν τα όρια της εσωτερικής αγοράς, έχουν παγκόσμια εμβέλεια. Γίνονται εργαλείο για βιομηχανική πολιτική και πολιτική καινοτομιών σε παγκόσμιο προσκήνιο για να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Καλωσορίζουμε τον εντοπισμό πέντε προτεραιοτήτων για τον τομέα της πληροφορικής που έχουν εντοπιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευφυής και αποτελεσματική χρήση της ενέργειας ε, και τα σωστά πρότυπα για τις μεταφορές, για ευφυή χρήση των ε, μεταφορών. Η DG Connect και η DG Growth θα πρέπει να συνεργαστούν επί κοινών πρωτοβουλειών για την πληροφορική μαζί με άλλους τομείς της βιομηχανίας που δεν σχετίζονται ε, με την πληροφορική για να αποφύγουμε μονομένες προσπάθειες και αλληλεπικαλύψεις. Η επιτυχία της βιομηχανίας μας εξαρτάται επί αποτελεσματικής ψηφιοποίησης. Άρα, χρειάζεται συμμετοχή στη διαδικασία τυποποίησης. Τα, αυτά τα πρότυπα θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τεχνολογία εχμής. Θα πρέπει να υπάρχουν σωστές σχέσεις μεταξύ έρευνας και ενοτομίας και θα πρέπει να προβλέψουν ανάγκες διαλειτουργικότητας. Πρέπει να έχουμε πρότυπα που ανταποκρίνονται στην τεχνολογική πρόοδο. Μεγαλύτερη εναρμόνιση απαιτείται σε ε, σχέσεις με τη ΣΥΠΑ για ε, τη χρήση του νέφους, υπολογισμού, ε, υπολογισμού νέφους και την ασφάλεια. θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντατικοποιήσει τη συνεργασία της με τρίτες χώρες όσον αφορά την τυποποίηση αυτή. Έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε τις, ευρω... τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες, να μπορούμε να πωλήσουμε πιο εύκολα τα ευρωπαϊκά προϊόντα στο παγκόσμιο, στην παγκόσμια αγορά. Αυτά είχα να πω, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σιγητά, η κυρία Σπυράκη, εκ μέρους της ομάδας του ΕΛΚ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χένκελ, για την πρώτη σας αυτή παρέμβαση. Προσβλέπω στο σχέδιο γνωμοδοτήσεως του κ. Χένκελ και την έκθεση ΙΜΚΟ για να έχουμε μια πιο συγκεκριμένη βάση για τις εργασίες μας. Εν τω μεταξύ, να εκφράσω κάποιες σκέψεις για τον εξυγχρονισμό των ευρωπαϊκών προτύπων βάσει της ανακοινώσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής του περασμένου Ιουνίου. Γιατί και πώς μπορούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω την ευρωπαϊκή τυποποίηση, το ESS, ε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησεως. Η απάντηση στο ερώτημα Ποια είναι. Εμεί είμαστε μέλη τη Επιτροπή Ήτρε για να υποστηρίξουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία, για να προσαρμοστεί ταχύτερα δυνατόν στι προκλήσει και τα προβλήματα. Αυτό είναι υποφελέ για του καταναλωτέ, των επιχειρηματιών, για του επιχειρηματίε και του εργοδότε. Αναβαθμίζοντα το ESS, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τύπο πίσω, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μα. Να σα δώσω κάποιου αριθμού από την ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Επίτροπη. Λοιπόν, ο αντίκτυπος της ανάπτυξης τυποποίησης εκτιμάται στο 0,8% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 0, για τη Γαλλία, 0,3% για το Ηνωμένο Βασίλειο και 0,9% για τη Γερμανία. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να μειώσουμε τον κατακαιρματισμό της ψυχιακής αγοράς. Συμφωνούμε νομίζω, καταρχάς, επ' αυτού. Ε, πρέπει να εξασφαλίσουμε και κάτι άλλο, για λειτουργικότητα των τεχνολογιών. Κάτι πολύ σημαντικό για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Άρα πρέπει να πετύχουμε μεγαλύτερο συντονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να προωθήσουμε ευρωπαϊκά πρότυπα, να μειώσουμε τα εμπόδια, να τάρουμε τα εμπόδια που προέρχονται από τον κατοικερματισμό. Άρα προσβλέπω συνεργασία μου τον κύριο Χένκελ. Και νομίζω ότι τελικά η γνωμοδότησή μας θα είναι πολύ ποιοτική. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Γκρίφιν, εκ μέρου των Σοσιαλιστών, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι κρίσιμο για τους πολίτες μας να βελτιώσουμε την εναρμόνιση των προτύπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι παρέχουν μεγαλύτερη προστασία για τους καταναλωτές, μεγαλύτερη σαφήνεια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μειώνει και το κόστος σε αυτή την υποποίηση. Η εναρμόνιση των ευρωπαϊκών προτύπων είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να πετύχει προτεραιότητά τη σε διάφορους τομείς που ανέφεραν οι συνάδελφοι. Και την ψυχιακή ενιαία αγορά, την ενεργειακή ένωση και να έχουμε πιο ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά Τώρα όσον αφορά την ψηφιακή ενή αγορά, το διαδίκτυο των αντικειμένων και το διαδίκτυο για τον κόσμο, για τον άνθρωπο, θα απαιτήσει εναρμονισμένα πρότυπα, αν θέλουμε να είναι κάτι εποφελές για τους Ευρωπαίους πολίτες. Η φύση της ευφυούς τεχνολογίας απαιτεί διασυνοριακή διασύνδεση. Παραδείγματο χάρη δεν υπάρχει αγορά για ευφύ αυτοκίνητα αν λειτουργούν μόνο τα αυτοκίνητα στα δικά μας ε, κράτη-μέλη. Είναι επίση αδύνατο να πετύχουμε του στόχου για την Ενεργειακή Ένωση χωρί να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα τυποποιημένα πρότυπα. Θα έχουμε καλύτερα περιβαλλοντικά πρότυπα, θα προωθήσουμε την καινοτομία με αυτόν τον τρόπο, θα έχουμε διαλειτουργικότητα μεταξύ δικτύων για την αύξηση της χρήση ανανεσίμων πηγών ενεργείας στο ενεργειακό μείγμα, χωρί να αυξήσουμε το κόστο για του χρήστε. Προσβλέπω στη συνεργασία με τους συναδέλφους μου επί του σημαντικού αυτού χαρτοφυλακίου και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Η κυρία Βαν Νόιβελχόιζε έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι περιμένω πώς και πώς τη συνεργασία με τον κύριο Χένκελ, τον εισηγητή, και τη συνεργασία με τους συναδέλφους, τους κοιόδης εισηγητές. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Συμφωνώ με τα προαναφερθέντα από τους συναδέλφους. Χωρίς σωστά πρότυπα δεν θα έχουμε εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς δεν θα έχουμε καν αγορά και δεν θα υπάρχει και διαλειτουργικότητα. Και αυτό είναι κάτι που διακαώς επιθυμούμε. Όλοι συμφωνούμε από αυτό. Ίσως να προβώ σε κάποια σχόλια σχετικά με το τι θεωρούμε σημαντικό για τη θέσπιση των προτύπων. Στην Επιτροπή ΕΚΟΝ έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο όσον αφορά την, ασφάλ... την ασφάλεια των προϊόντων. Πρέπει να είναι τυποποιημένα και ασφαλή και απλά. Μιλάμε για τυποποίηση, αλλά απλά προϊόντα και διαφάνεια, και αυτές οι λέξεις είναι σημαντικές, και νομίζω ότι θα πρέπει να εστιαστούμε επ' αυτού. Αν θέλουμε να θεσπίσουμε τα πρότυπα, θα πρέπει αυτά τα στοιχεία να τα λάβουμε υπόψη που ανέφερα. Να είναι σαφή, ξεκάθαρα, απλά, στο βαθμό του δυνατού. Δεύτερον, καινοτομία, νέα τεχνολογία, Κινείται πολύ γρήγορα η τεχνολογία. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να επιταχύνουμε τη διαδικασία καθορισμού προτύπων. Επίσης συμφωνώ με αυτό που ήδη είπε και ο Σχένκελ. Δηλαδή, θα πρέπει επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στον καθορισμό των προτύπων. Όχι μόνο διότι θα δεχτούν πιο εύκολα έτσι τα πρότυπα αυτά και στις διαγραφές, αλλά έτσι θα πετύχουμε και καλύτερα πρότυπα πρότυπα τα οποία πραγματικά θα μπορούν καθημερινά να εφαρμόζονται και να λειτουργούν και να δίνουν αποτελέσματα. Τέλος, ε, να τονίσω ότι θα πρέπει διατομιακά να καθοριστούν τα πρότυπα. Το είπε και η συνάδελφος από τους σοσιαλιστές. Ο τομέας της ψηφιοποίησης με το διαδίκτυο των αντικειμένων ε, έχουμε διάφορους τομείς πολιτικής που ενώνονται και δεν πρέπει να είναι απομονωμένοι και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Χρειάζεται διατομεακή προσέγγιση. Και τέλει συμφωνώ με τα αναφερθέντα, δηλαδή ότι είναι υπέροχα τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά διεθνή πρότυπα είναι ακόμα καλύτερα. Αν μπορέσουμε να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση και αυτό θα ήταν πάρα πολύ επικοδομητικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Νίον Χόιζα που μίλησε εκ μέρους του ECR, εκ μέρους του Ισάλτε. Άλτε. Μην κάνουμε λάθη, μην κάνουμε λάθη. Όχι, όχι, όχι, λέει ο πρόεδρο. Εκ μέρου τη Άλτε μιλήσατε. Ο εισηγητή είναι εκ μέρου του ΙΣΙΑΡ. Ζητώ συγγνώμη. Αλλά έτσι είχα τη δυνατότητα και εγώ να προφέρω σωστά το όνομά σα. Νιούενχάουζα. Πάντα μου αρέσει, πάντα μου αρέσει να κάνω αυτό, κύριε πρόεδρε. Εκ μέρου τη Γκουε, ο κύριο Σιλικιώτη έχει το λόγο. Ε, ε, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χέγγελ και να πω ότι αναμένω ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία. Ε, για την ομάδα μας στην Ευρωπαϊκή Νοτική Αριστερά είναι ξεκάθαρο πως η έκθεση της Επιτροπής όσον αφορά την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών προτύπων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του 21ου αιώνα πρέπει να θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο να έχει ως βασικό γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών και των συμφρόντων της κοινωνίας των καταναλωτών αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δυστυχώ σήμερα τα ευρωπαϊκά πρότυπα αποτελούν μια διαδικασία τυποποίηση που εξυπηρετεί το στόχο για δημιουργία και ενίσχυση της ενιαίας αγοράς προωθώντας κυρίως την ανταγωνιστικότητα ε, και έχει ως αποτέλεσμα αυτοί που αποφελούνται από τα ευρωπαϊκά πρότυπα να είναι κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις και ε, οι πολυεθνικές. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή πρέπει να έχουμε στόχο να πετύχουμε ευρωπαϊκά πρότυπα που να εξυπηρετούν πραγματικά την κοινωνία, να οδηγώντα την άπτυξη νέων ποιοτικών θέσεων εργασία, ενισχύοντα τα πρότυπα ασφάλεια και ποιότητα, στηρίζοντα την πραγματική οικονομία ε, και ένα από του στόχου είναι να προωθήσουμε ε, μέσω τη καινοτομία και τη έρευνα την επαναβιομηχανοποίηση ε, ιδιαίτερα σε περιοχές κυρίως του Νότου. Ε, εξίσου σημαντικό είναι να ασφαλίσουμε πως τα ευρωπαϊκά πρότυπα ε, δεν πρέπει να λειτουργούν σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά θα τις στηρίζουν ώστε να μπορούν αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η, τεράστια πλειοψηφία ε, των επιχειρήσεων στην Ευρώπη και είναι ο, ο βασικός άξονας της οικονομίας της Ευρώπης ε, να τις βοηθούν για να ε, αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και τις καινοτόμους μεθόδους. Ε, τέλος, στη διαδικασία ανάπτυξη των ευρωπαϊκών προτύπων είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια επικοδομητική συνεργασία, να ληφθούν υπόψει όλων των κοινωνικών εταίρων, ιδιαίτερα των συνδέσμων καταναλωτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, αλλά και των τοπικών κοινοτήτων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ πολύ, λέει και ο Πρόεδρος. Η κυρία Κάπελ από το ΕΕΝΕΦ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα κοινά πρότυπα όταν πρόκειται για την ε, καινοτομία και είναι απαραίτητο να συμβάλλουν αυτά τα πρότυπα έχει ήδη αναφέρει ο, ο εισηγητής την σημασία αυτή για την πληροφορική και γενικά για την ε, παροχή υπηρεσιών. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια ψηφιοποιημένη αγορά και το ανέφερε αυτό η διοσηγητής ότι η νεφόδης υπολογιστική ε, διαδικασία είναι πάρα πολύ σημαντική για να δώσει στην ε, ε, βιομηχανία τις δυνατότητες να είναι ανταγωνιστική. Επίσης και η, τα πρότυπα για τον τομέα παροχής υπηρεσιών. 70% της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι αυτή τη στιγμή μέσα στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών και επομένω είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να έχουμε τα κατάλληλα πρότυπα και στον τομέα αυτό. Τα πρότυπα οδηγούν σε περισσότερη καινοτομία και τα πρότυπα <clears throat> μπορούν με τον τρόπο αυτό να προκαλέσουν περισσότερη οικονομική ανάπτυξη και τόνωση της απασχόλησης. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες καταδεικνύουν ότι τα πρότυπα έχουν πολύ θετικέ επιπτώσεις για την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Μπορούν να προσθέσουν περίπου 0,9% σε οικονομική ανάπτυξη και υπολογίζεται σε 17 δισεκατομμύρια ευρώ η εξοικονόμηση η οποία μπορεί να προκύψει από καλύτερη χρήση των πρότυπων. Όλα αυτά είναι σημαντικά στοιχεία και έτσι μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία μπορεί να ενσωματωθεί καλύτερα και η ευρωπαϊκή οικονομία. <clears throat> Είναι λοιπόν και νέες αγορές οι οποίες μπορούν να κατακτηθούν χάρη στα πρότυπα αυτά. Αυτό μας επιτρέπει να μειώσουμε το κόστος αλλά συγχρόνως να αυξήσουμε την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων. <clears throat> Είναι σημαντικό εδώ να λαμβάνονται υπόψη και οι θέσεις των εμπλεκομένων έχει γίνει και στο παρελθόν, αλλά είναι απαραίτητο να γίνεται με πιο ταχύ ρυθμό, γιατί γίνονται πιο ραγδαία οι εξελίξει και είναι απαραίτητο για να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μα να υπάρχει τακτική επικαιροποίηση των προτύπων σε συνεργασία και με τρίτες χώρες ώστε τα ευρωπαϊκά πρότυπα να μπορούν να γίνουν παγκόσμια πρότυπα και αυτό θα μπορέσει να διατηρήσει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Ευχαριστώ, Λέω ο Πρόεδρος. και από την Ευρωπαϊκή Κομισιόν ο διευθυντής της DigiGrow η κυρία Κέλστεν Γιόρνα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για τα πρότυπα η Κομισιόν θέλει να έχει μια στενή συνεργασία με το Συμβούλιο αλλά και το Κοινοβούλιο. Είναι μια από τις καινοτομίες που έχουμε στο πακέτο μέτρων που παρουσιάζουμε στις 19, παρουσιάσαμε στις 19 Απριλίου και την 1η Ιουνίου εφέτος. Εδώ η καινοτομία είναι ότι θα παρουσιάζουμε κάθε χρόνο μια διαθεσμική έκθεση στα άλλα θεσμικά όργανα πριν από την έγκριση του προγράμματος εργασίας για τα πρότυπα που πρέπει να υποβάλει κάθε χρόνο τον Ιούλιο η Κομισιόν επί τη βάση του κανονισμού για τα πρότυπα του 2012. Ξέρουμε βέβαια τον χρονισμό της έκθεσής σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποβάλουμε την εγκαίρωση την έκθεσή μας στη διαθεσμική ως συμβολή στη συζήτησή σας. Η έκθεση αυτή θα δώσει την δυνατότητα για όλα τα θεσμικά όργανα να κάνουν ένα απολογισμό της προόδου που έχει επιτευχθεί, να εξετάσουν τις τρέχουσες πρωτοβουλίες και να διακριβώσει τις ανάγκες οι οποίες πρέπει να εξυπηρετηθούν από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προς όφελος των εταιριών μας και των πολιτών μας. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. <clears throat> Ξαναγυρίζω στις τελευταίες αυτές ε, παρατηρήσεις που μπορεί να μας δώσει ο κ. Χέγγελ, ο εισηγητής για να κλείσουμε τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ έχω περάσει όλη την επιχειρησιακή μου ζωή στον τομέα αυτό από την εποχή των διάτριτων δελτίων έως το διαδίκτυο και πάντα γκρίνιαζα στον εαυτό μου και στους συναδέλφους μου για το επίπεδο των προτύπων στην Ευρώπη με τις συμβολές των σκιωδών συναδέλφων μου καθώς και με τις προτάσεις που διατυπώνονται από την Κομισιόν, έχω μεγάλες προσδοκίες ότι θα μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί για να κλείσουμε αυτό το χάσμα και να φτάσουμε πιο κοντά σε μια ψηφιακή ενιαία αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Το χρονοδιάγραμμα τώρα <clears throat> είναι ακόμα η υποδιαπραγμάτευση με την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς που είναι η αρμόδια επί της ύλης και προβλέπουμε να υπάρχει μια, πρωτο... μια προθεσμία για τις τροπολογίες μεταξύ 17 και 19 Ιανουαρίου. 12 με 17 Ιανουαρίου μάλλον λέει ο πρόεδρος. Θα έχουμε τότε <clears throat> ένα έγγραφο βέβαια στην Επιτροπή μας γιατί η σημερινή συζήτηση ήταν απλώς μια ανταλλαγή απόψεων με δίχως έγγραφο. Θα έχουμε μια περαιτέρω συζήτηση στις 12 και 17 ε, Ιανουαρίου πριν από την εκπνοή της προθεσμίας για τις τροπολογίες. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο στην μέση διάταξή μας, το σημείο 5, η αντιμετώπιση του γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακρίσεων που οφείλονται στην υπηκότητα των τόπων κατοικίας και των τόπων εγκατάσταση των πελατών εντό τη εσωτερική αγορά. θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων και δίνω καταρχήν το λόγο στην εισηγητρία μας, την κυρία Εύα Καϊλή η οποία εκπροσωπεί την Επιτροπή μας και έρχεται από την Σοσιαλιστική Ομάδα. Έρχεται το λόγο κυρία Καϊλή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, τους τελευταίους μήνες έχω εξεργαστεί αυτή την πρόταση κανονισμού <clears throat> που αφορά τον γεωγραφικό αποκλεισμό και άλλες μορφές διακρίσεων που έχουν να κάνουν με την υπηκοότητα, την ηθαγένεια ή τον τρόπο διαμονής των πελατών. Η πρόταση της Κομισιόν νομίζω ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και αποτελεί τμήμα ενός φιλόδοξου πακέτου για να διευκολύνει το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι πάντα μια μεγάλη πρόκληση για μας ως Επιτροπή Ήτρε. Πρέπει να εξασφαλίσουμε μια εξισορροπημένη προσέγγιση, λαμβάνοντα υπόψη τα συμφέροντα των καταναλωτών, αλλά και των παραγωγών και εμπόρων. Είναι απαραίτητο λοιπόν να αντιμετωπίσουμε και τα εμπόδια και τους φραγμούς που μπορούν να οδηγήσουν σε διακρίσεις, όταν οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν να έχουν <clears throat> μια υπηρεσία ή ένα αγαθό που βρίσκεται σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να τα λαμβάνουμε αυτά υπόψη. Ο στόχος του κανονισμού είναι να εξασφαλίσει ότι μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε, αγαθά με προσβάσιμο τίμημα και έτσι να προωθήσει τον ανταγωνισμό. Δεν είναι ο χώρος που θα πρέπει να οδηγήσει σε αλλαγή των κανόνων για τα οπτικοακουστικά και το copyright. Ο στόχος είναι να υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση των πολίτη σε υπηρεσίες ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του θέση. Και έτσι στο παρελθόν η μετακίνηση από μία ιστοσελίδα σε μια άλλη θα γίνεται ε, αυτόματα, θα έχει πάντα τη δυνατότητα ο πολίτης να επανέλθει στην αρχική του επιλογή. Επομένως θα τελειώσει αυτή η ματαιωτική πρακτική, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επομισθούν δυσβάσταχτο κόστος και θα μπορέσουν να διατηρήσουν την ελευθερία του επιχειρήν. Η υποχρέωση λοιπόν αυτή που πρέπει να επιβληθεί δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι ο πάροχος ή ο πολιτής θα πρέπει να είναι υποχρεωμένος να παραδώσει ένα προϊόν εκτός του τόπου όπου λειτουργεί. Και επίσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν επιχειρησιακές τακτικές που επιλέγουν όσο δεν κάνουν διακρίσεις ε, εναντίον ορισμένων καταναλωτών. Δεν θέλουμε λοιπόν να έχουμε ένα υπερβολικό γραφειοκρατικό άγχο σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η συμμόρφωση με τον κανονισμό δεν θα σημαίνει υποχρέωση κάλυψης ή θα σημαίνει την ανάγκη να πάρουν πίσω ένα προϊόν σε ορισμένε περιπτώσει. Και αυτό δεν θα πρέπει να οδηγεί προβλήματα εφόσον δεν υπάρχει διαμεθοριακή παροχή ενός προϊόντος, ο νόμος καταναλωτών της χώρας είναι αυτός ο οποίος ισχύει και για τις πληρωμές. Θα πρέπει να γίνεται δεκτή μια πληρωμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανεξάρτητα από τη χώρα από την οποία εκείνη. Αυτό θα δώσει δυνατότητα στους καταναλωτές να αγοράσουν προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τον κίνδυνο να μην είναι δεκτή η πληρωμή. Στο παρελθόν, ορισμένοι καταναλωτές δεν είχαν πρόσβαση σε αγαθά αλλά και υπηρεσίε λόγω της πηγής της διαδικασίας πληρωμών. <clears throat> Επίσης, θα πρέπει να μειωθούν και τα τέλη που επιβάλλουν οι εταιρείε πιστοτικών καρτών βάσει της αντίστοιχης ομιλίας για να μπορέσουν να διευκολυνθεί και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Περιμένουμε λοιπόν να υπάρχουν απλώς τα ελάχιστα απαραίτητα τέλη με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις συναφείς συναλλαγές θα πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχει συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρχει προστασία των δεδομένων που θα αποδικεύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει επίση να έχουμε νομοθεσία η οποία θα είναι αποτελεσματική και φιλική προς τον χρήστη. Είναι απαραίτητο λοιπόν να λάβουμε υπόψη όλα τα στοιχεία τα οποία μπορούν να περιληφθούν σε αυτό το νομοθέτημα. Το copyright και άλλα στοιχεία δεν εμπίπτουν σε, αυτήν την, σε αυτό το νομοθέτημα. Το θέμα λοιπόν της ε, μεταφοράς οπτικού ακουστικού υλικού είναι κάτι το οποίο εξετάζεται σε άλλα νομοθετήματα. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να δώσουμε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση στον καταναλωτή και μια φιλικότερη προς την επιχείρηση προσέγγιση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι είναι πράγματι ένα βήμα προς μια ε, φιλική προς το χρήστη επιγραμμική αγορά στην Ευρώπη και μπορεί να είναι μια βάση για άλλες σημαντικές αποφάσεις όπως η μεταρρύθμιση του οπτικοακουστικού και του copyright επίσης την καταγραφή ΦΠΑ, είναι κάποιες από τις αποφάσεις που θα πρέπει να κάνουμε προς την σωστή κατεύθυνση και νομίζω ότι αυτά όλα είναι θετικά. Θα πρέπει να ισχύουν και οι ίδιες αρχές πάντα, το να είμαστε φιλικοί προς τον καταναλωτή αλλά και προς, την, προς τους παρόχους. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία σας αυτή. Ίσκυρωτης τώρα, Herbert Royal πρώτα που αντικαθιστά την κυρία Νίμπλερ εκ μέρου του ΕΡΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να φύγω βέβαια, δεν μπορώ να παραμείνω πολύ περισσότερο, έχω μια συνάντηση. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και θα ήθελα να τονίσω ότι ο στόχος αυτού του νομοθετήματος είναι να μπορεί ο καταναλωτής να έχει επιγραμμική πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες σε μια άλλη χώρα χωρίς καμία διάκριση. Επομένως θα πρέπει να βελτιωθεί η διαδικασία ε, εμπορίου προϊόντων αυτού του είδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα εμβαθύνει και θα ενισχύσει την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι και λογικό και ε, χρήσιμο. Θα πρέπει λοιπόν να πάψουν να υπάρχουν στεγανά στον τομέα αυτό και επίσης πρέπει να κάνουμε τα απαραίτητα να μπορούν να βρεθούν λογικές και πρακτικές λύσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να θέλουν να παραμείνουν μονάχα σε περιφερειακές αγορές και δεν θα δραστηριοποιηθούν κατά ανάγκη στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ε, είναι καλό ότι δεν λαμβάνονται υπόψη σε αυτή τη στιγμή τα, οι οπτικοακουστικές πτυχές, γιατί υπάρχουν και σημεία τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν χωριστά. Η Αγγέλικα Νίμπλερ μου, είπε να εκφράσω την προσδοκία της ότι αυτά τα οποία θα γίνουν μέσα στα πλαίσια αυτού του νομοθετήματος δεν θα πρέπει να επηρεάσουν καθόλου την επιχειρηματική δυνατότητα ε, επιλογής και την ελευθερία του επιχειρήν είναι, κάποιο στοιχείο το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη σε όλες τις περιπτώσεις και είπαμε ότι ορισμένα στοιχεία όπως το οπτικό, ακουστικό ή το copyright δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την ε, περίπτωση και φυσικά επίσης δεν θέλουμε να επηρεάσουμε την αδότητα των επιχειρηματιών να καθορίζουν το τίμημα α, των υπηρεσιών. Η Αγγέλικα Νίμπλερ θα είναι παρούσα στι μεταγενέστερε διαβουλεύσει, αλλά αυτέ είναι οι πρώτε σκέψει που ήθελα να σα δώσει. Ευχαριστούμε πολύ. ECR. Τώρα, ο κύριος Τονονεύσκη, που είναι σκιώδης εισηγητής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Καϊλή για το σχέδιο εκθεσής της. Μπορώ να συμφωνήσω με πολλά από αυτά που είπε και συμφωνώ επίσης γενικά με τα λόγια της. Συμμερίζω λοιπόν κάποια σχόλια από πλευρά τη ομάδα μου. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι ο αδικαιολόγητος γεωγραφικός αποκλεισμός, ή διακρίσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν, πρέπει να καταργηθούν, έτσι ώστε να μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε την ενιαία αγορά. Δεν πρέπει να δημιουργούνται εμπόδια χωρίς λόγο. Μερικές φορές όμως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί μερικές φορές οι καταστάσεις είναι περίπλοκες. Δεν θα πρέπει να επιφέρουμε διοικητικό άχθος και θα πρέπει να μην παρεμβαίνουμε σε αγορές οι οποίες ήδη λειτουργούν καλά. Συμφωνώ λοιπόν ότι δεν πρέπει να υπάρχει υποχρέωση και συμφωνώ επίσης ότι δεν πρέπει να υπάρχει υποχρέωση να παίρνει κανείς πίσω ε, παραδόσεις. Αυτά είναι πράγματα τα οποία κάνουν πιο δύσκολη τη ζωή για τους εμπορευόμενους. Συμφωνώ επίσης ότι η ελευθερία η σύμβασης πρέπει να γίνεται σεβαστή. Δεν πρέπει να υπάρχουν ειδικά σώματα που θα δημιουργηθούν για αυτόν εδώ το σκοπό. Κάτι άλλο με το οποίο μπορώ να συμφωνήσω είναι ότι πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει η μεταρρύθμιση για το copyright και ίσως να συζητηθεί τότε. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ όλους τους κοιόδης συζητητές. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Βέρνικ, εκ μέρους της Άλντε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Καηλή, την εισηγήτρια, για την ε, παρουσίασή της. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι υπάρχει δυνατότητα και μπορούμε να υποφεληθούμε με καλύτερη διασύνδεση στην αγορά μας. Είναι κάτι που πρέπει να γίνεται σε θελοντική βάση, αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω για την οικονομία μας, την επιγραμμική, την online. Άρα, ο γεωγραφικός αποκλισμός που περιορίζει αυτήν την αγορά πρέπει να πάψει να υπάρχει όταν είναι δικαιολόγητος. Θέλουμε λοιπόν να αρθούν τα εμπόδια τα οποία παραμένουν στην εσωτερική μας αγορά. Είναι δύσκολο μερικές φορές να αγοράζουν οι πολίτες προϊόντα από άλλες χώρες ή να κυκλοφορήσουν προϊόντα μιας επιχείρησης σε όλες τις χώρες. Ο γεωγραφικός αποκλεισμός όμως δεν είναι και το μόνο εμπόδιο για να έχουμε μια νέα ψηφιακή αγορά. Υπάρχουν και διάφορες εθνικές προδιαγραφές που διαφέρουν μεταξύ τους το κόστος της μεταφοράς αλλά και άλλες διαφορές στην εθνική νομοθεσία. Για την ανακύκλωση για παράδειγμα. Και όλα αυτά τα ζητήματα επίσης πρέπει να κάνουμε κάτι. Τώρα, για την ε, πρόταση αυτή πιστεύουμε ότι έχει πολλά θετικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα συμφωνώ ότι ο αγοραστής δεν πρέπει να είναι θύμα διακρίσεων εξαιτίας της γεωγραφικής του θέσης ή της υπηκότητάς του. Δεν ε, πρέπει όμως να υπάρχει υποχρέωση. Θα είναι τεράστιο βάρος αυτό για τις επιχειρήσεις μας και κυρίως για τις ε, μικρές επιχειρήσεις που εμπορεύονται στο ίντερνετ. Έπειτα είναι πολύ σημαντικό ο καταναλωτής να δίνει την άδειά του κάθε φορά που ε, στέλνει ο αρχικός εμπορευόμενος στο διαδίκτυο, τον καταναλωτή, σε μια άλλη διεύθυνση. Επίσης δεν πρέπει να υπάρχει διάκριση για τις πληρωμές που γίνονται online. Χωρίς αυτά τα στοιχεία η πρόταση αυτή θα αποτελεί κοινό γράμμα, κοινό και θα παραμείνει ο γεωγραφικός αποκλεισμός. Υπάρχουν ε, και διάφορα θέματα τα οποία πρέπει να υπογραμμιστούν ακόμα περισσότερο. Για μένα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι σε αγορές όπου δεν είναι ενεργός ο εμπορευόμενος, αλλά υπάρχει μόνο παθητική στάση, τότε θα πρέπει να είναι η χώρα η οποία αποφασίζει για το τι θα ισχύει. Οι εμπορευόμενοι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν όσο γίνεται μεγαλύτερη ελευθερία σε μια συμβατική σχέση και χωρίς την ψηφιακή αγορά. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι προσβλέπω σε καλή συνεργασία με την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές για να καταλήξουμε σε μια ξεκάθαρη γνωμοδότηση της Επιτροπής μας η οποία θα δώσει περισσότερα κίνητρα και καλύτερη κατάσταση στην εσωτερική μας αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, μία Πρόεδρος. Ο κύριος Τσόκα, ΕΝΕΦ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, καλημέρα συνάδελφοι. Ευχαριστώ την εισηγήτρια την κυρία Καηλή. Ο κανονισμός αντιμετωπίζει πολύ ενδιαφέροντα θέματα και πολύ επίκαιρα και εμπεριέχει και σημεία με τα οποία συμφωνούμε. Όμως για να συμβάλλουμε και με κριτική προσέγγιση αλλά επικοδομητικά διότι θέλουμε όλοι μαζί να κάνουμε τα αναγκαία και να έχουμε νομοθέτημα τόσο ώστε να έχουμε και το σωστό, να υπάρχει και το σωστό θάρρο να χρησιμοποιείται τελικά αυτό το νομοθέτημα. Για να το κάνουμε αυτό, η πρόταση κανονισμού θα πρέπει σε κάποια σημεία να να έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Έτσι, όπως διατυπώνεται, να φέρεται στα αίτια της διαφοροποιημένης προσέγγισης στην αγορά που οφείλεται κυρίως στον κατακαιρματισμό όσον αφορά την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδείγματο χάρη, για να δώσουμε κάποια παραδείγματα, οι εθνικές νομοθεσίες διαφέρουν για την ετικετοθεσία, για την πιστοποίηση, ε, διαφορετικό κόστος της εργασίας και θα μπορούσαμε να δώσουμε πάρα πολλά άλλα παραδείγματα που είναι αίτια που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως αίτια και θα πρέπει να τα σκεφτούμε αυτά μην αντιμετωπίζετε στα πραγματικά αίτια τις ρίζες που εμποδίζουν πελάτες και επιχειρήσεις να αγοράζουν και να πουλούν αγαθά και υπηρεσίες έξω τα σύνορα, με την πρόταση του κανονισμού ως διατυπώνεται δεν μπορούμε να καταφέρουμε να είμαστε αποτελεσματικοί όσον αφορά την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διασυνοριακής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι σημαντικό λοιπόν κατά τη διάρκεια των εργασιών μας να λάβουμε υπόψη κατά ταπεινή μου άποψη, τη σημαντική συνεισφορά που ήδη έχει γίνει 433 απαντήσεις Φερρυπίν που κατέθασαν όσον αφορά το νομοθέτημα από τους καταναλωτές, από επιχειρήσεις, από ενώσεις και από κράτη-μέλη που σίγουρα θα είναι σημαντικά σημεία να ληφθούν υπόψη διότι αυτοί οι εμπλεκόμενοι φορείς ε, αντιπροσωπεύουν τον πραγματικό κόσμο και πιστεύω ότι ο νομοθέτης μπορεί να κάνει καλή δουλειά αν ξεκινήσει κάτωθεν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Άλλοι ομιλητέ τώρα. Η κυρία Κάλλας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ε, καλή δουλειά που έχει γίνει για την έκθεση αυτή. Το νομικό πλαίσιο πρέπει να είναι σαφές για τους εμπορευόμενους. Και όταν πρόκειται για παθητικές πωλήσει, γιατί δεν είναι σαφή τα όρια. Η γεωγραφική, ο γεωγραφικός αποκλεισμός σημαίνει ότι όταν κάποιος δεν πουλάει σε μια χώρα, τότε δεν μπορούν να εφαρμοστούν στις πωλήσει αυτές και οι νόμοι της χώρας. Προσεφωνώ με την πρόταση της εισηγήτριας που διακρίνει στους τρόπους πληρωμής. Έχουμε ενίο χώρο πληρωμών, διασφαλίζεται η ασφάλεια των πληρωμών, οπότε πρέπει να μην χρειάζεται καν να ρωτάμε κατά πόσο δικαιολογείται η διάκριση. Για τις πληρωμές Θέλω επίσης να υπογραμμίσω και τη διάκριση που γίνεται με τις πληρωμές που μερικές φορές απαιτούν ένα τηλέφωνο σε κάποιες χώρες μέλη για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Είναι κάτι το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει παραβλέψει. Και τέλος, νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε και το εύρος εφαρμογής το πεδίο εφαρμογή. Το παράδειγμα των μεταφορών που αποκλείεται, αλλά δεν θα έπρεπε να αποκλείεται από το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Εγώ δεν καταλαβαίνω την αιτιολόγηση. Εδώ υπάρχει ο γεωγραφικός αποκλεισμό, το copyright κτλ. Αν όμως περιορίσουμε το πεδίο εφαρμογής τόσο πολύ, τελικά δεν μένει και τίποτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Ο κ. Σον Κέλλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Εύα και τους κοιόδης ηγητές για τις προτάσεις τους. Εν γέννη είναι καλά ισορροπημένες οι προτάσεις. Θα μας βοηθήσουν ούτω ώστε να πετύχουμε τη φιλοδοξία μας. Να ολοκληρώσουμε την ψηφιακή ενιαία αγορά κατά τη διάρκεια της θητείας μας και κυρίως να επιστρέψουμε να επιτρέψουμε την ευημερία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πάντα κουβεντιάζουμε για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Πρέπει να άρουμε του περισσότερου φραγμού που μπορούμε όσον αφορά την εύρυθμη λειτουργία του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτό αυτή. Και ο γεωγραφικό αποκλεισμό, το geo-blocking, είναι ένα από του φραγμού ο οποίο θα πρέπει να ε, αρθεί. Όπω είπαν κάποιοι ομιλητέ, πρέπει να προσέξουμε. Να μην υπερβάλλουμε και σε κάποιε περιπτώσει θα πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες. Άρσος δυνατότητας πώληση και επιβίωση ενδεχομένως για κάποιους εμπλεκομένους φορείς. Ας πούμε, να μπορούν αθλητικά σωματεία να απολούν τα τηλεοπτικά της δικαιώματα, τα διφωνικά δικτά κλπ. στο εξωτερικό. Ένας φορέας του οποίου προείδρευα στην Ιρλανδία αθλητικός σύνδεσμος πολλούς δικαιώματα σε διάφορους εξωτερικούς ε, φορείς για εκπομπές στην Ευρώπη. Πρέπει, θέλουμε φιλελευθερωποιημένη αγορά, αλλά πρέπει να βρούμε σωστή ισορροπία. Αν το πετύχουμε αυτό, θα είναι σημαντικότατη εξέλιξη. Και έτσι θα ολοκληρωθεί η ενιαία ψηφιακή αγορά. Θα πλησιάσει η ολοκλήρωση. Ευχαριστώ την Εύα και τους συναδέλφους και προσβλέπω σε περαιτέρω συζητήσεις μαζί τους και να προχωρήσουμε σε αυτόν τον τομέα. Αυτά και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Αγαπητέ συνάδελφοι, ευχαριστούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. κύριος Βέρνερ Στέγκ, επικεφαλής της μονάδας ε, της Γενικής του DG Connect. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Δεν έχω να πω πολλά. Εν γέννη συμφωνώ με όσα άκουσα στην αίθουσα. Ευχαριστώ πολύ τους ομιλητές. άκρος επικοδομητική προσέγγιση. Όλα αυτά τα σημεία που θίξατε είναι σχετικά εν συγκρίση με το στόχο της προτάσεως. Θέλουμε να πετύχουμε σωστή ισορροπία. Θέμα ισορροπίας είναι εδώ μεταξύ θεμητών επιθυμιών και συμφερόντων καταναλωτών και εξίσου θεμητά συμφέροντα εμπορευομένων κυρίως μικρών επιχειρήσεων. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε. Μη δικαιολογημένε διακρίσει να με καταπολεμήσουμε. Αυτό είναι το βασικό. Όπω είπαν πολλοί ομιλητέ, πάντα υπάρχουν λόγοι για του οποίου οι έμποροι δεν θέλουν να πωλήσουν σε άλλα κράτη-μέλη. Θέλουμε να απομονώσουμε κάποιε περιπτώσει όπου θεωρήσαμε ότι το κόστο και το κίνδυνο για του εμπορευομένου όταν, όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με κάποιες υποχρεώσεις ήταν πολύ ε, περιορισμένοι κίνδυνοι, αν υπήρχαν καν. Και αυτό σχετίζεται με αυτά που είπαν, μη διασυνοριακή παράδοση, που είναι πολύ δαπανηρή. Τίποτα στην προτάση δεν ζητά εναρμόνιση των τιμών. Οι έμποροι μπορούν να προσφέρουν διαφορετικέ τιμέ σε διαφορετικέ αγορέ προφανώ. Όταν ο καταναλωτή πηγαίνει σε μια συγκεκριμένη στοσελίδα δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διάκριση. Θέλουμε να προστατεύσουμε τι υποχρεώσει μετά πώληση. Το είπε η κυρία Καϊλή. Τα αγαθά που δεν δίδεται στην αγορά άλλου κράτους μέλους. Επίσης, παθητικές πωλήσει και δεν υπάρχει κατεύθυνση δραστηριοτήτων προς άλλες επικράτειες, αν δεν κάνει τίποτα άλλο για να κατευθύνει δραστηριότητε του, Ποιες είναι οι ευθύνε του εμπορευόμενου, ποιο νόμο ισχύει. Από ό,τι είδα τι τροπολογίε σα, όλε οι τροπολογίε ακολουθούν την κατεύθυνση διευκρινήσεω των σημείων αυτών. Και αυτό είναι κάτι πρόσδεκτο. Πνευματικά δικαιώματα των οπτικοακουστικών μέσων, όπως αναφέρθηκε, είναι ε, σε ξεχωριστό πεδίο. Στη μεταρρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων. Το όλο πεδίο εφαρμογή του κανονισμού ευθυγραμμίστηκε με την οδηγία υπηρεσιών. Και αυτό για πολύ σωστού λόγους η οδηγία αυτή υπηρεσιών εξαιρεί τι οπτικοακουστικέ υπηρεσίε. Αναφέρθηκε ότι δεν ασχολούμεθα με τι ρίζε του προβλήματο, του κατακαιρματισμού, ανέφερε ο Ιταλό συνάδελφο. Πράγματι, δεν έχουν αυτό σκοπό τα μέτρα. Συμπληρώνουμε εδώ τα διάφορα άλλα μέτρα που προτάθηκαν για την ψηφιακή ενία αγορά και για το ηλεκτρονικό εμπόριο για να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά εμπόδια. Εδώ, εν τη απουσία πλήρους εναρμονίσεως, υπάρχουν μεν πολλά εμπόδια που απομένουν, όμως προσπαθούμε να δώσουμε μεγαλύτερη επιλογή και στον ε, καταναλωτή την μια μεριά και μεγαλύτερη ασφάλεια στον εμπορευόμενο για τις πληρωμές. Αυτό που ε, είπε η κυρία Κάλλας, βασιστήκαμε στο κεκτημένο των χρηματοσυντικών υπηρεσιών. Δεν ξεπερνάμε αυτό το όριο αλλά βασιστήκαμε σε αυτά στον κανονισμό συναλλαγών και λοιπά και διάφορους κανονισμούς και βασιζόμαστε επιφυσταμένων κανόνων και υποχρεώσεων. Σκοπός να περιορίσουμε το κόστος και το κίνδυνο για τους εμπόρους, για το κεκτημένο χρηματοστατικών υπηρεσιών, όπως είπατε μερικοί από εσά, εισάγει το θέμα ταυτοποίησης του καταναλωτού για να καλύπτεται και ο έμπορος αν κάποιος ε, πελάτης πάει να πληρώσει με πλαστά μέσα πληρωμής. Μπορώ εδώ να σταματήσω πιστεύω, διότι δεν άκουσα κάτι με το οποίο να διαφωνώ και να έπρεπε να διαμαρτυρηθώ. Ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στη συνέχιση των συζητήσεων με την Επιτροπή. Ευχαριστώ, Λεοπρόεδρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας και τώρα η εισηγήτριά μας, η κυρία Εύα Καηλή, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα επικοδομητικά σας σχόλια. Ήδη ε, βοήθησαν τα σχόλιά σας, αλλά προσβλέπω ε, στις τροπολογίες σας. Έχουμε ακόμα χρόνο και για άλλες τροπολογίες. Είναι σημαντικό επίσης σαν ήτρα να καταλήξουμε σε κοινή θέση που αντιπροσωπεύει τη λογική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, λαμβάνοντα υπόψη του καταναλωτέ τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ευρωπαϊκή οικονομία αν δεν μιλάμε για πλήρη εναρμόνιση, όμως θα γίνουν πολλές μεταρρυθμίσεις, ένα κομμάτι των μεταρρυθμίσεων που θα γίνουν. Άρα αποτελεί αυτό που κάνουμε ένα κομμάτι άλλων εκθέσεων που θα ετοιμάσουμε. Να επαναλάβω ότι αυτή η πρόταση είναι ένα βήμα προς τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο διαδίκτυο φιλικό προς το χρήστη. Αλλά θέλουμε επίσης να πάρουμε αποφάσεις πιο πέρα. Μεταρρύθμιση του πνευματικού δικαιωμάτος στις του υπηρεσίες, παράδοση πακέτων ε, και άλλα θέματα τα οποία πρέπει να καλύψουμε για να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον φιλικό προς τους χρήστες και τις επιχειρήσεις, μια πραγματικά ενιαία ψηφιακή αγορά και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία μου. Για τα σχόλιά σας και για την σύνοψη της συζήτησης. Και τώρα η προθεσμία τροπολογιών είναι η επόμενη Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου. Έχουμε μερικές μέρες ακόμα λοιπόν, <clears throat> μέχρι το μεσημέρι λοιπόν της 14 Νοεμβρίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή μας στις 12 Ιανουαρίου. Και στην ε, ΙΜΚΟ που είναι η αρμόδια Πετσίλης στις 25 Απριλίου λέει ο πρόεδρος. Αυτό είναι το χρονοδιαγράμμά μας. Λοιπόν, ευχαριστώ για τη συζήτηση, αγαπητοί τώρα συνάδελφοι. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο, το σημείο υπαριθμών 6, ενημέρωση σε σχέση με τις ενεξελίξεις διαπραγματεύσεις για την ενεργειακή επισήμανση. Ο κύριος Ταμπουράνο είναι ο εισηγητής μας και το σύστημα εμπορίας εκπομπών με τον κύριο Φέδερ, λέει. Ο κύριος Ταμπουράνο μου έστειλε ένα σχέδιο της ομιλίας του, διότι δεν μπορούσε να έρθει. Θα διαβάσω λοιπόν αυτά που λέει. Και εγώ να πάρω σε ένα τμήμα των διαπραγματεύσεων. Μπορώ να δώσω και κάποιες προσωπικές παρατηρήσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Λοιπόν, η ενεργειακή επισήμανση. Μέχρι τώρα έχουμε λάβει χώρα τρεις τριγωνικοί διάλογοι. Μέσα Ιουλίου, αρχές Σεπτεμβρίου και τέλος της 11 Οκτωβρίου του 2016. Μέσα σε υψηλού επίπεδου διαθεσμική ανταλλαγή απόψεων με την Προεδρία, ο Υπουργός Ιβαν Κορτσόκ και με την ε, συνέλευση των Προέδρων, το Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε την ε, στεναρή του στάση για το άρθρο 12, δηλαδή κατ' εξουσιοδότηση πράξης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην ε, συζήτησή μας και έχουμε τρία σημαντικά σημεία σε ό,τι αφορά την ενεργειακή επισήμανση. Τρία κύρια σημεία. Ένα από αυτά είναι η κατεξουσιοδότηση των εφαρμοστικών πράξεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζει ο κ. Ταμπουράνο έχει περατώσει ένα πακέτο αντιπροτάσεων που περιλαμβάνει και το άρθρο 7, αλλαγή κλίμακο που παρουσιάστηκε στις 11 Οκτωβρίου και το άρθρο 11 που αφορά την βάση δεδομένων και το παράτημα 1 που αφορά τα δεδομένα στις 20 Οκτωβρίου 2016 και έχει παρουσιάσει επίσημα τις προτάσεις αυτές στην Προεδρία. Δύο σημαντικά θέματα, η ανα αλλαγή κλίμακος της ε, τράπεζα και η τράπεζα δεδομένων. Αυτά είναι θέματα να εξελίξει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει κατ' επανάληψη την στεναρή του θέληση να σεβαστεί την δέσμευσή του για την επίτευξη μιας συμφωνίας για το σύνολο κανονισμό υπό Σλοβακική Προεδρία. Υπογραμμίζω και εγώ το ίδιο, το υπογράμμισα το ίδιο όταν συναντήθηκα με την Κορεπέρ, του εκπροσώπους των κρατών μελών, πριν από λίγες εβδομάδες. Το επόμενο σημείο στο γράμμα του κ. Ταμποράνα, αν ευδοκιμήσουν όπως ελπίζω <clears throat> οι τρέχουσες προσπάθειες, ο τέταρτος τριγωνικός διάλογος θα μπορούσε να λάβει χώρα τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου 2016, αλλιώς θα πρέπει να γίνει στις αρχές του 2017 υπό Μαλτέζικη Προεδρία. Έρχομαι λοιπόν τώρα στα τρία πιο σημαντικά σημεία. Η αλλαγή κλίμακος. Έχει προχωρήσει εκεί πέρα η διαπραγμάτευση και επετεύθη μια συμφωνία για όλα τα στοιχεία εκτός από δύο. Γενικά το χρονοδιάγραμμα το οποίο πρέπει να τύχει σεβασμού για την <clears throat> αλλαγή ταξινόμησης των ετικετών αφορά τρεις κατηγορίες, ταχεία, μέση και βραδία. Επομένως, αυτά αφορούν το χρονοδιάγραμμα και τέλος. Η απόλυξη η οποία πρέπει να επιλεγεί <clears throat> μέσα στη διαδικασία αυτή αλλαγής της κλίμακος Και τώρα πάμε στη βάση δεδομένων. Εκεί είναι ακόμα πιο προχωρημένη συζήτηση. Έχει υπάρξει συμφωνία για όλα τα μείζωνα θέματα με την εξαίρεση του λεπτομεριακού καταλόγου τεχνικής τεκμηρίωσης και τον κεντρικό τομέα της ε, συμμόρφωσης για το πρόγραμμα και επίσης για τις τους τρόπους που θα χρησιμοποιήσουν οι αρχές εποπτείας της αγοράς για να ζητήσουν από τους παραγωγούς περαιτέρω τεχνική τεκμηρίωση η οποία μπορεί να είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και τρίτον η διευκρίνηση τυχών επικαλύψεων ώστε να αποφευχθούν αυτές. Αυτά λοιπόν τα τρία σημεία που δεν είναι πολύ εύκολο να καλυφθούν, αλλά αυτά είναι το περιεχόμενο τη επιστολής του κυρίου Ταμπουράν και το μεγάλο σημείο υπαριθμό 3 είναι ότι ο φάκελος αυτός περιλαμβάνει και ένα σημαντικό στοιχείο διαθεσμικού χαρακτήρα. Η επιλογή κατεξουσιοδότηση ή εφαρμοστικών πράξεων. Όπως ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα δημοκρατικού ελέγχου στις κάτι εξουσιοδότηση πράξεις που του δίνει το δικαίωμα κυρία Στις εφαρμοστικές πράξεις όμως δεν μπορούμε να τις κάνουμε τίποτα, ούτε καν να τις ακυρώσουμε. Η τωρινή οδηγία για την ενεργειακή ε, αποδόση και την σήμανσή της, καθώς και η πρόταση της Κομισιόν, η νέα πρόταση λοιπόν που συζητούμε τώρα, και οι δύο αμφί προβλέπουν την χρήση κατεξιοδότηση πράξεων. Αυτή είναι και η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει την πρόταση της Κομισιόν προ την κατεύθυνση αυτή, γιατί αυτό βασίζεται στο τωρινό πλαίσιο, το οποίο λειτουργεί πολύ καλά. Αλλά αντιθέτω το Συμβούλιο ακολουθώντας την πάγια πρακτική του από τον Νοέμβριο του 2015, έχει μετατρέψει όλες τις κατεξουδιώτες πράξεις σε εφαρμοστικές πράξεις, το οποίο σημαίνει ότι αποστερεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το δικαίωμά του να <clears throat> θέσει εμπόδια στις ρυθμίσεις βάσει κανονισμού. Δεδομένου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν κάνει μια διαθεσμική συμφωνία πριν από λίγους μήνε για την καλύτερη νομοθεσία όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμπεφώνησε να υπάρχουν παράγοντε εμπειρογνώμονες των κρατών μελών κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής πράξης, φάσης μάλλον των κατεξουσιοδότηση πράξεων, έχουμε μια νέα λύση και ενδεχομένως θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε στην βράχυνση της προπαρασκευαστικής περίοδου. Αλλά δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο ακόμα. Κάποια από αυτά που είπα ήταν και η δική μου εμπειρία. Το πιο σημαντικό είναι ότι στον τελευταίο τριγωνικό διάλογο και σε συνάντηση με τον πρέσβη Μικόφτσιν της Σλοβακικής Προεδρίας και με τους κορεπεράδες όλων των κρατών μελών πριν από ένα μήνα έκανα ιδιαίτερα σαφές το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να δεχτεί την πρόταση του Συμβουλίου για τη μετατροπή των κατεξουσιοδότηση πράξεων σε εφαρμοστικές, Όσα έχει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Έχουμε εδώ πολλούς, πολλά επιχειρήματα, το ιστορικό, την πρόταση της Κομισιόν, τη δυνατότητα παρουσίας των εμπειρογνωμόνων κατά τη διάρκεια της προπαρασκευής κάθε εξουσιοδότηση πράξεων και την βράχυνση της χρονικής διάρκειας της προετοιμασίας. Οι ισχυώδεις ηγητές θα συναντηθούν αργότερα σήμερα να συζητήσουν το θέμα αυτό εν ώψη των ε, αλλαγών που έχουν γίνει το τελευταίο μήνα <clears throat> με στόχο να περατωθεί αυτό το νομοθέτημα υπό Σλοβακική Προεδρία. Αλλιώς θα αναλάβει τη σκητάλη η Μάλτα. Θα είναι όμως καλύτερο να μπορέσει να τελειώσει μέσα στην Σλοβακική Προεδρία αυτή η διαδικασία. Αυτά. Θέλουν να προσθέσουν κάτι οι σκιώδεις εισηγητές, γιατί ο εισηγητής μας δεν είναι παρόν. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, οι σκιώδεις. Κύριε Ρόιλ, θέλετε να πείτε κάτι. Όχι, λέει ο κύριος Ρόιλ. Η κυρία Βέρινγκ, από την άλλη. Όχι, νομίζω ότι τα είπατε πολύ ξεκάθαρα και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you, colleagues. So. Ευχαριστώ αυτοί οι συνάδελφοι. Επομένως, αυτό αφορούσε την ενεργειακή επισήμανση, τον πρώτο τρίλογο. όπου αρμόδιος ο κ. Σταμπουράνο. Έχουμε τώρα το σύστημα εμπορίας εκπομπών με τον Φρεντερίκο Φέντερλεϊ, ο οποίος είναι επικεφαλής. Βέβαια, θα πρέπει να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας, αλλά προηγουμένως θα πρέπει να γίνει και συζήτηση και ψηφοφορία στην Επιτροπή Ένβη. Θέλουμε λοιπόν να δούμε πώς αντιμετωπίζεται το θέμα αυτό από την Επιτροπή αυτή και αν μπορώ να ζητήσω από τον κύριο Φέντερ λέει, να μας δώσει μια έκθεση για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Όπως όλοι γνωρίζετε, η ψηφοφορία έλαβε χώρα 13 Οκτωβρίου και μπορέσαμε να έχουμε ευρεία ε, στήριξη στη δικιά μας θέση. Και μάλιστα ευρύτερη στη ψηφοφορία από ό,τι είχα φανταστεί αρχικά. Το αποτέλεσμα μου δίνει σαφή εντολή για να εκπροσωπήσω την άποψη της έντρη και στην συνάντηση με τους σκιώδες στην ΕΝΒΗ. Πράγμα που κάνω. Είναι σαφές για μένα ότι η ομάδα της Επιτροπής Περιβάλλοντος ε, κοιτάζει με αρκετή όρεξη την ε, τοποθέτηση της Ήτρε. Υπάρχουν ε, διάφορες συμβαστικέ προτάσεις του εισηγητή που βασίζονται στη γνωμοδότηση τη δικιά μας. Φυσικά υπάρχουν σημαντικά ζητήματα πάνω στα οποία πρέπει ακόμα να δουλέψουμε. Η συνάντηση με τους σκιώδεις εισηγητές πάντως στην ΕΝΒΗ κατέληξε με προτάσεις συμβιβαστικές όσον αφορά την αναλογία ανάμεσα στην αγορά και την, την εκτός, ο περίφημος διακανονισμός Duncan, και μπορέσαμε να έχουμε κάποια βάση συμβαστική. Δεν λέω ότι έχουμε καταλήξει, αλλά στη συζήτηση πάντως ε, ελήφθη υπόψη σοβαρά η άποψη της Ήτρε και συζητήθηκε και θα ληφθεί υπόψη και στη συνέχεια των συζητήσεων. Υπάρχουν κάποια σημεία που άλλαξαν σήμερα για τα κονδύλια που έχουμε επιμερισμένη ευθύνη και εμείς. Είναι ένα νέο ζήτημα για την ομάδα της ΣΥΤΡΕ. Εγώ θα μιλήσω με τους δικούς μας σκιώδεις και την πλειοψηφία. ΕΛΚ, ECR, ε, ΑΛΔΕ, να είμαστε έτοιμοι για το πώς πρέπει να κινηθούμε στη συνέχεια των διαπραγματεύσεων. Παραμένουμε ομάδα Ήτρε λοιπόν στις διαπραγματεύσεις που έχουμε με την ΕΝΒΗ. Προσπαθώ να είμαι και επικοδομητικός και να εξισορροπήσω καλά τις συζητήσεις κάθε φορά που υπάρχει ένα διέξοδο στην ΕΝΒΗ, προτείνω τη θέση της Ήτρε σαν συμβιβασμό και διέξοδο. Εννοείται ότι πρέπει να πετύχουμε ευρία συνένεση όχι μόνο στην Επιτροπή μας αλλά και στο, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, τι θα γίνει αν δεν ε, τελειώσουμε θετικά. Θα πρέπει να υπάρξει τριμερής διάλογος. Εγώ θα συζητήσω με τους Γιώδης και ανάλογα με το αποτέλεσμα θα δούμε αν η δικιά μας θέση έχει ληφθεί επαρκώς υπόψη ή όχι. Και ανάλογα θα αποφασίσουμε τη συνέχεια. Οι πλειοψηφίε φαίνονται κάπως διαφορετικές στην Ήτρε και στην Ένβη. Και ποιος ξέρει και στην Ολομέλεια. Από την άλλη, αν οι δύο επιτροπές έχουν ε, μεταξύ τους συνοχή, θα μπορέσουμε πιο εύκολα να προχωρήσουμε σε τριμερή διάλογο. Πάντως είναι καλό που συζητάμε και που πρότεινα και εγώ μια μεθοδολογία και θα βάλουμε και θέματα εμείς ως ομάδα Ήτρε βάσει των όσων μου λένε και οι συνάδελφοι και θα τα συζητήσουμε στην ΕΝΔΕ. Εξακολουθούν να παραμένουν εκκρεμότητες, πρέπει να το πω. Οπότε μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Μέχρι τώρα Πάντως η δικιά μας η άποψη γίνεται σεβαστή και έχει ληφθεί υπόψη σε πολλές σεβαστικές προτάσεις της ΕΝΒΗ. Αυτή είναι η κατάσταση. Είχαμε τρεις συναντήσεις με τους Κιώδης και σήμερα μία και αρχίζουμε να μπαίνουμε στην ουσία. Και χαίρομαι που το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν τόσο ξεκάθαρο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Έτσι μπορούμε να τηρήσουμε και το χρονοδιάγραμμα. Αν είχαμε αργήσει, τότε δεν θα είχα σαφή εντολή από την Επιτροπή μας για να ξέρω προς τα που πρέπει να κινηθώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε για τόσα μας είπατε. Ξέρουμε ότι κάνατε πολύ σκληρή δουλειά και στις πολιτικές μας ομάδες το ξέρουμε ότι οι σκιώδες συζητητές μας δούλεψαν σκληρά. Είναι καλό να συμμεριζόμαστε τις ίδιες απόψεις με την ΕΝΒΗ. Ο κύριος Ρούμπικ τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον εισηγητή. Νομίζω ότι είναι εξισορροπημένη πρόταση που παρουσιάζει στην Επιτροπή μας την Ήτρε και καλύπτει τα συμφέροντα όλων των πλευρών με ορθό τρόπο πιστεύω. Και αυτός θα πρέπει να είναι και ο στόχος να καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη πρόταση, να αποφύγουμε τη μετακίνηση επιχειρήσεων και θέσεων απασχόλησης, διότι δεν πρέπει να ενισχύσουμε περισσότερο την ανεργία στην Ευρώπη. Θα πρέπει να διατηρήσουμε και τις επενδύσεις στην Ευρώπη και όχι να φύγουν από την Ευρώπη και η καινοτομία να παραμείνει και αν θέλουμε να έχουμε μια ισχυρή, ένα ισχυρό κοινωνικό ιστό χρειαζόμαστε μια στεναρή και εύρωστη βιομηχανία και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μια επαναβιομηχάνηση, όχι μόνο με 20% της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας μέχρι το 2020, που είναι ένα στόχος που δεν έχουμε πετύχει, αλλά θα πρέπει να φτάσουμε στο 30% του ΑΕΠ στην, στην δευτερογενή παραγωγή στη βιομηχανία. Έτσι μπορούμε να έχουμε περισσότερες θέσεις απασχόλησης και ενίσχυση του κοινωνικού ιστού. Γι' αυτό θα πρέπει να διαπραγματευτούμε και πάλι με την ε, Envy, τα... οι πρόσοδοι που έρχονται από το σύστημα ETS θα πρέπει να τεθούν στην υπηρεσία του εξυγχρονισμού, ώστε να μπορέσουμε με τον τρόπο αυτό να προσελκύσουμε νέε επενδύσει και να δημιουργήσουμε νέε θέσει απασχόληση. Τα χρήματα αυτά δεν θα πρέπει να πάνε στην κατανάλωση, αλλά θα πρέπει να αποδοθούν σε επενδύσεις για να επιτύχουμε τους στόχους μείωση των εκπομπών. Αν <clears throat> λοιπόν όλο και περισσότερο μειώνεται ο ρόλος της Ευρώπης στα θέματα αυτά, θα έχουμε περισσότερα προβλήματα. Σας παρακαλώ λοιπόν το ταμείο αυτό του εξυγχρονισμού να δημιουργηθεί, γιατί είναι μια από τις βασικές μας διεκδικήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι και στο, στην Ολομέλεια όταν έρθει το θέμα αυτό είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί ώστε να έχουμε την ευκαιρία οι όλοι οι βουλευτές να εκφράσουν την άποψή τους ώστε με τις ενεργές μας να μην αυξήσουμε, να μην οδηγήσουμε σε αύξηση την ε, ανεργία, αλλά αντίθετα να δημιουργήσουμε καλές θέσεις στο εργασίας και να προστατεύσουμε και το περιβάλλον με υποδειγματικό τρόπο στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Ανίμπλερ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ μπορώ να συμφωνήσω απόλυτα με αυτά τα οποία λέει ο κύριος Ρούμπιν και εγώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εισηγητή για την πλήρη πληροφόρηση που μας έδωσε σε σχέση με την τωρινή κατάσταση των διαπραγματεύσεων στον τομέα αυτό της εμπορίας των εκπομπών. Θα ήθελα λοιπόν <clears throat> να επιμείνω ότι θα πρέπει να υπερασπιστούμε τη θέση της Επιτροπής Ήτρε έναντι της Επιτροπής Ένβη. Ο κύριος ε, Φέντελε έχει κάνει μια εξαιρετική εργασία. Αναφέρθηκε στο θέμα αυτό και ο κύριος Ρούμπι και εσείς κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζουμε ότι υπήρξε η ανάγκη να συζητήσουμε διαμακρών για τα θέματα αυτά και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να προασπίσουμε τη θέση της Ευρωπαϊκής ε, της ε, Επιτροπής Ήτρε και αυτό σημαίνει και μια ευρωπαϊκή προοπτική για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, να παραμείνουν οι βιομηχανίε σε μας και να μην υπάρξει μετακίνηση επιχειρήσεων και να χαθούν θέσεις εργασίας, να χαθεί η έρευνα και η ανάπτυξη, να... και έτσι να μειωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, θα πρέπει λοιπόν να τα διατηρήσουμε όλα αυτά και να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία μεταξύ αυτών που κάνουμε εμείς για τη μείωση των εκπομπών και αυτών που γίνονται από άλλες χώρες του κόσμου. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το γεγονός ότι είχατε ένα ανοιχτό πνεύμα για να ακούσετε τις απόψεις όλων των ε, πολιτικών ομάδων. Ευχαριστώ λοιπόν και για τον τρόπο με τον οποίο διενεργήσατε τις διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό. Για την περαιτέρω τώρα διαδικασία και εγώ συμφωνώ. Όλα αυτά εξαρτώνται από το αποτέλεσμα το οποίο θα προκύψει από και την Επιτροπή Ένβη και μετά θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε αν δεν μας ικανοποιεί η θέση της ε, Επιτροπής Ένβη. Θα πρέπει να περάσουμε σε περαιτέρω αλλαγές πρώτου φτάσουμε στην Ολομέλεια. Είναι χρήσιμο να μπορέσουμε να έχουμε μια εκ νέου συζήτηση και συντονισμό μεταξύ μας ώστε να δώσουμε το ειδικό βάρος και την στεναρότητα της θέσης του Κοινοβουλίου που είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το Συμβούλιο. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να αφήσουμε μόνο μια πλειοψηφία στην να αποφασίσει και εμείς προηγουμένως θα πρέπει να τα προετοιμάσουμε στην Επιτροπή μας. Ο κύριος Ρόελ. Ευχαριστώ Ρόελ. Πάρα πολύ σύντομα. Εγώ βρίσκω σωστή την πρόταση του κύριου Φέντελε ότι πρέπει να προχωρήσουμε με ταχαία βήματα. Βέβαια θα πρέπει να έχουμε μια σωστή στάση. Νομίζω ότι η... ήταν δύσκολη η διαδικασία να βρούμε κάποια ε, ισορροπία σε σχέση με τα πιστοποιητικά εκπομπών τα οποία αγοράζουν οι επιχειρήσεις και αυτών τα οποία δίδονται χωρίς τίμημα σε επιχειρήσεις. Νομίζω ότι σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να φτάσουμε σε μια ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Όταν έχουμε ένα τόσο σημαντικό θέμα δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει μονάχα από τις αρμόδιες επιτροπές. Είναι και θέμα δημοκρατίας και πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε στο τέλος να ε, να φτάσουμε σε μια ο, ψηφοφορία στην Ολομέλεια για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να προσθέσω με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι προλίγου ότι πετύχαμε τελικά συμβιβασμό μετά από μακροσκελέστατες συζητήσεις στην Επιτροπή Ήτρε. Είναι πολύ ισορροπημένο συμβιβασμός μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Μεγάλη επιτυχία αυτή η δική σας Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Συζητήσαμε το θέμα διότι θέλαμε μάλιστα να σας ενθαρρύνουμε να διατηρήσετε τη θέση της Επιτροπής μας. Είμαστε βέβαιοι ότι είσαστε πεπισμένος για τη θέση μας. Είστε πεπισμένος γι' αυτή, αλλά θα θέλαμε να σας ενθαρρύνουμε. Διότι κάποιοι από εμά ήμασταν μέλη της Επιτροπής ΕΝΒΗ, ξέρουμε ότι η ατμόσφαιρα εκεί είναι πολύ διαφορετική από ό,τι εδώ. Σας καταλαβαίνουμε απόλυτα. Καμιά φορά ήταν δύσκολα τα πράγματα. Και ήταν θέμα ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Είναι κανόνας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτός. Σαν συνήθεια θα έλεγα. Και όχι τόσο σαν κανόνας. οι συνδεδεμένε αυτές οι επιτροπέ βάσει του άρθρου 54, αν κινούμεθα σε αυτό το πλαίσιο, καταλήγουμε στην ε, Ολομέλεια. Δεν είναι κάτι γραμμένο. Συνήθως αυτό κάνουμε. Δυνάμει του άθρου 54, μάλλον πρέπει να πάμε στην Ολομέλεια, διότι στις ψηφοφορίες στην Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς τι θα γίνει. Αν μας καλύπτει ή δεν μας καλύπτει η θέση εκεί που ψηφίζεται ή όχι. Πολύ καλύτερα θα ήταν να πούμε ότι η τελική ψηφοφορία θα πρέπει να λάβει χώρα στην Ολομέλεια ε, για να δοθεί εντολή από το Ευρωκοινοβούλιο για τη διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ εκ νέου για την προσέγγισή σας και για τα αστηριότητά σας. Εισηγητά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους Ρούμπιχ, Νίμπλερ, Ρόιλ και εσάς κύριε Μπούζεκ, κύριε Πρόεδρε, ε, για τα καλά σας λόγια. Πρέπει ε, Επίσης να ευχαριστήσουμε και τους Κιώδης και τα τέσσερα κόμματα που συμμετέχουμε. Επανέλαβα πάντα στις διαπραγματεύσεις ότι πρέπει να υπάρχει βούληση ε, και το αποτέλεσμα να είναι κάτι που δέχονται όλοι. Ε, να είναι κάτι εύπεπτο ούτως ή πίν. Δεν είναι πάντα εύκολο αυτό. Και αυτός είναι ο σκοπός του συμβιβασμού είναι λίγο δυνηρός για όλους, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι πολύ πιο εύκολο και έτσι μπορούμε να πάμε στις ομάδες μας και να πούμε, κοιτάξτε, ε, συμβάλαμε σε αυτό το αποτέλεσμα μέσω του συμβιβασμού. Αν σταθούν οι ομάδε ότι δεν συνέβαλαν σε συμβιβασμό, τότε ποιο ο λόγος να έχουμε ένα συμβιβασμό. Αυτό είναι το ένα. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σα. Συμφωνούν οι σκιώδει. Αν μπορώ να πω ποια είναι η αποψή του για αυτά που είπατε, θα γίνουν διαβουλεύσει την επόμενη εβδομάδα. Ξέρω ότι η δουλειά μου από πλευρά φιλελευθέρων ολοκληρώθηκε. Ε, μετά την ψηφοφορία σαν εισηγητής ε, πρέπει να φροντίσω να περάσει η θέση αυτή μέσω της ψήφου της πλειοψηφία. Το έχω αναλάβει αυτό και θα προσπαθήσω να προωθήσω τη θέση μας και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Θα συνεχιστεί η δουλειά, θα συνεχιστεί ο διάλογος με τις τέσσερις ομάδες που ε, συνυπογράφουν ε, τις συμβαστικές αυτές λύσεις. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ κύριε Σιγητά, ευχαριστώ Φρέντερικ. Ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο. Πάμε στο σημείο 7. Επίσκεψη στο Κάλαρας 24 Οκτωβρίου. Ενημέρωση. Συνάδελφε Όγγεν Φλόιντ, Κλάρ Μούντι, Μύροσλαβ Πόχε και ο Φλάβιος Σαβονάτο. Τέσσερις συνάδελφοι, λοιπόν. Είναι να ξεκινήσουμε ο καθένας με τη σειρά του. Συνάδελφε Φρόιντ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να εκφράσω την πίκρα μου και την απογοήτευσή μου εξ αρχής. Θα συζητήσουμε το θέμα της πιο περίπλοκης προωθημένης τεχνολογίας που έχουμε επισκεφθεί ποτέ. Και εδώ είμαι και έχω το στικάκι μου με ένα βίντεο της επίσκεψής μας όπου κινηματογράφησα κάθε μέρος που επισκεφθήκαμε και τα πάντα όσα μπορούσαμε να δούμε και μου είπαν ότι είναι αδύνατον να τρέξω αυτό το βίντεο τον 21ο αιώνα σε αυτή την αίθουσα. Αυτό είναι το κενό που πρέπει να ξεπεράσουμε όταν μιλάμε για την ε, τεχνολογία. Θα ακούσατε, κύριε Πρόεδρε, ότι θα ξεκινούσα την παρουσίασή μου και τη συζήτησή μου βάσει του βίντεο λέγοντας ότι θα μιλήσουμε για τη μεγαλύτερη μηχανή καύσης χρημάτων ε, ή τον σωτήρα της ανθρωπότητας. Αυτό είναι το ίτερ. Η αντιπροσωπεία μας πήγε στο ίτερ στις 24 Οκτωβρίου τα μέλη της αντιπροσωπείας αναφέρατε κάποιους από αυτούς, θα προσέθετα τον Κρίστιαν Άιλερ, τον Φλάβιο Τζανονάτο, τον Τζάκομ Νταλούντε από τους Πράσινους που ήταν μεταξύ εκείνων που έπρεπε να αναφερθούν. Συναντηθήκαμε με τον Μπενάν Μπικό, τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Φορέα Ήτρε, τον Γιονχάνες Βέμπερ, εκτελεστικό διευθυντή της Σύνδεξης για Ενέργεια, της υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη για το Ήτρε, Ήτερ ε, μάλλον πέρασαν χρόνο μαζί μας, μας εξήγησαν τις περίπλοκες λεπτομέρειες ε, του πειραματικού αντιδραστήρα. Αν όλα λειτουργήσουν, αν τα πάντα λειτουργήσουν, αναμένεται το ΙΤΕΡ να δείξει ότι είναι εφικτό να ε, παράξουμε ενέργεια της τη σύνδεξη για ελληνικού σκοπούς. Θα παράξουμε άφθονη, ασφαλή, καθαρή και οικονομική φθηνή ενέργεια, αν πετύχει. Έχουμε τρία προβλήματα βασικά τεχνολογικό πρόβλημα κατασκευής του τόκαμακ, δηλαδή του πυρήνα του αντιδραστήρα. Η πρόκληση είναι να βάλουμε όλα τα τμήματα που πρέπει και πώς να διαχειριστούμε τη διεθνή συνεργασία. Εδώ μιλάμε για ένα πρόγραμμα που είναι κοινό μεταξύ Ευρώπης, Κίνας, Ινδίας, Ιαπωνίας, Κορέας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ευρώπη πληρώνει περίπου 45% του εφοδιασμού και οι άλλοι πληρώνουν ο κάθε εταίρος περίπου 9% ο καθένας. Όπως ξέρουμε ε, η πολυμερής προσέγγιση είναι κάτι υπέροχο θεωρητικά. Στην πράξη όμως ε, μπορεί να γίνει κάτι αρκετά άκαμπτο. Για το ίτερ σημαίνει ότι επί σειρά ετών το έργο αυτό δεν ακολούθησε σωστή πορεία χρειαστήκαμε και άλλο ένα σχέδιο δράσης που ετοιμάστηκε το 2015 για να καθορίσουμε σαφείς προτεραιότητες και χρονοδιάγραμμα για τις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις. Αυτά τα βήματα προόδου συμπεριλαμβάνουν τη θέσπιση διαδικασίας λήψης αποφάσεων και ελέγχου. Ο Γενικός Διευθυντής Μπιγκό έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις. Πρέπει να καθορίσουμε ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για τη λειτουργία και τη χρήση πλάσματος μέχρι το 2025 αντί του πρώτου στόχου που ήταν το 2020 και να παράξουμε ισχύ το 2035 από σύνδεξη. Άρα δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το δούμε αυτό. Εσείς και εγώ. Ελπίζουμε, ελπίζω και ελπίζω και για σας και εσείς να το δείτε τότε. Να εκτεμήσουμε καλύτερα τους αναγκαίους πόρους για να πετύχουμε το χρονοδιάγραμμα πρέπει να έχουμε σωστά βήματα καθορίσουμε για την απόδοση. Αυτά είναι τα βήματα προόδου τα οποία θα πρέπει να επιτευχθούν. Πρέπει να γίνεται ανεξάρτητη αποτίμηση του προγράμματος, βελτίωση με αυτή την αποτίμηση της λειτουργής προγράμματος και το ευρωπαϊκό τμήμα, η σύνδεξη για παραγωγή ενέργειας, ε, είναι υπεύθυνο για τρία βήματα. Πρώτα απ' όλα το πρόγραμμα ITER στο Κανταράς που επισκεφθήκαμε, Δεύτερον, συνεργασία με την Ιαπωνία επί τριών προγραμμάτων έργων για τη σύνδεξη, ευρύτερη προσέγγιση όπως αποκαλείται, και τρίτον, η νέα γενιά των πειραματικών αντιδραστήριων σύνδεξης. Συνεργαζόμαστε με διάφορες φορείς, εταιρείες κλπ. για να κατασκευάσουμε τα ανταλλακτικά για το ίτερ και δημιουργούνται πολλές ευκαιρίες για τη βιομηχανία, για την έρευνα, ανάπτυξη, εργαστήρια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δημιουργούμε βιομηχανική βάση για σύνδεξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κλείνοντα να πω ότι η δομή διακυβέρνηση του ΙΤΕΡ και του προγράμματο σύνδεξη για ενέργεια είναι περιπλοκότατος μηχανισμός. Όπως είπα, αντιμετωπίστηκαν δυσκολίες, αλλά το έργο δίνει αποτελέσματα, είναι ορατό, μακάρι να μπορούσα να τα δείξω. Και συνεχίζεται η προσπάθεια. Επίσης, αυτό αφορά και τη σύνδεξη για παραγωγή ενεργείας. Θα σταματήσω εδώ και θα αφήσω τα λοιπά να τα πούνε οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ, με τρομάξατε συνάδελφοι που λέτε ότι αυτή η έρευνα δεν είναι για μένα, τι είπατε. Ότι, ότι θα τα δω με τα ματάκια από το 2035. Εντάξει, καλό είναι και το 2035, καλό μου φαίνεται. Θα τα καταφέρω. Ναι. Τέλειο και για μένα. Η κυρία Κλέρ Μούντι έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ναι, προφανώς όλοι προσβλέπουμε στο 2035. Ευχαριστώ τα σχόλια του κύριου Φρόιντ. Δεν ξέρω βέβαια τι κομμάτι έχει μείνει. Πάντως από αυτά που είδαμε και τα σχόλιά του θα συνεχίσουμε. Είναι όντως ένα εκπληκτικό πρόγραμμα και πραγματικά είναι πολύ κρίμα που δεν μπορούμε να δούμε το βίντεο που ετοίμασε ο συνάδελφος, γιατί είναι εκπληκτικό το τι έχουν πετύχει εκεί οι άνθρωποι. Αλλά δείχνει ακριβώ και τι μπορούμε να πετύχουμε παγκοσμίω όταν ασχολούμαστε με το θέμα της κλιματικής αλλαγής, γιατί περί αυτού πρόκειται. γίνεται ένα βήμα μπρο με τη συνθήκη του COP21 στο Παρίσι και εδώ είναι ένα ολόκληρο πρόγραμμα σε παγκόσμιο επίπεδο για να καταλήξουμε στις λύσεις που τόσο πολύ χρειαζόμαστε όσον αφορά τις ενεργειακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και την κλιματική αλλαγή. Αλλά και την ε, ασφάλεια στον εφοδιασμό ενέργειας. Δεν ήταν βέβαια ένα εύκολο πρόγραμμα, εννοείται δεν περιμένει κανείς να είναι εύκολο. Με τόσο πολύτιμους στόχους και τόσο δύσκολα ζητήματα επιστημονικά. Τώρα όμως υπάρχει. Με ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. Βάσει των αλλαγών στο πρόγραμμα δράσης του 2015. Από εκεί και πέρα υπάρχουν βήματα βάσει των οποίων μπορούμε να αξιολογήσουμε το πρόγραμμα, πόσο πετυχαίνει τους στόχους δηλαδή. Υπάρχει λογοδοσία και έλεγχος της διαδικασίας και από το εξωτερικό. Αλλά καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο ε, οικονομική συνεισφορά. Είναι και σε είδος ουσιαστικά από τις άλλες χώρες εκτός Ευρώπης. Ήθελα σχέση και με τις διαχειριστικές ε, αρχές των άλλων χωρών, αλλά είναι και θέμα της αλυσίδας εφοδιασμού για να είμαστε σίγουροι ότι αξιολογούμε σωστά όλα τα βήματα. Υπάρχουν βέβαια ζητήματα που έχουμε και πρέπει να έχουμε όσον αφορά τα επιτεύγματα αυτά του πλάσματος για το 2025, ώστε να πετύχουμε το στόχο που είπαμε πριν το 2035. Το θέμα των περιορισμών, τι μπορεί να πάει στραβά, τα πρόβλεπτα από τώρα μέχρι το 2025. αλλά όλα εξαρτώνται και από τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε για τον έλεγχο. Τέλος. Κάτι που αντικατοπτρίζει και αυτά που είπε ο Όρεγκον. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το όραμα αυτού του προγράμματος και το τι μπορεί να επιτευχθεί όχι μόνο στο τέλος που φυσικά είναι ζωτική σημασία στόχος, αλλά και το τι θα έχουμε μάθει κατά τη διάρκεια της εξέλιξης. Για αυτή την υπέροχη πηγή ενέργειας θα έχουμε μάθει για τα υλικά, για τη ρομποτική, τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ανάπτυξη τεχνολογίας υψηλής ποιότητας τόσο πολλές πίνο θα έρχονται από, αυτό το πρόγραμμα προκειμένου να πετύχουμε τον τελικό στόχο της σύνδεξης. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ όλους τους συναδέρφους. Φέτος είμαι συγητής για τους τελικούς λογαριασμούς κοινών ε, τέτοιων προγραμμάτων στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν εγώ έχω μια διαφορετική οπτική γωνία, έτσι, λογιστικού τύπου. Είναι ένα φοβερό πρόγραμμα τεχνολογικά μιλώντας και όχι μόνο. Και πρέπει να αναγνωρίσω ότι έχει επιτευχθεί τεράστια πρόοδος τους τελευταίους μήνες. Αυτό έγινε χάρη στην ε, νέα διαχείριση στην αδίκηση που άρχισε να λειτουργεί και έχουμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή νέα διαχείριση του προγράμματος αυτού. Έτσι λοιπόν, τώρα στεκόμαστε περισσότερο στα τεχνολογικά, στα κριτήρια τα οποία έχουν τεθεί και συνεργαζόμαστε καλά και με τους διεθνείς προμηθευτές. Δεν μπορεί παρά να είναι επιτυχία. Είναι λοιπόν σημαντικό να είμαστε και διπλωματικά ενεργοί στο Συμβούλιο της ΙΤΕΡ. Πρόκειται να γίνει συνεδρία σε σύντομα και θα είναι μια ευκαιρία να πετύχουμε παρετέρω πρόοδο. Κάποια πράγματα τα βλέπω εγώ κάπως διαφορετικά από τους συναδέλφους. Πρώτα από το οικονομικό ζήτημα το κόστος αυξάνει και υπάρχουν και καθυστερήσεις. Άρα δεν ξέρω αν θα πετύχουμε την προθεσμία του 2025. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο πρέπει να τα προσέξουν αυτά. Πάντως υπάρχουν κίνδυνοι, τους οποίους όμως δεν μπορούμε να περάσουμε. Εξωτερικοί κίνδυνοι, διεθνών σχέσεων. Στις διάφορες συζητήσεις που είχαμε στο κατω ρωτήσαμε πολλές φορές για τη σταθερότητα των εταίρων, είτε πρόκειται για την Ρωσία, είτε για το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit. Και σήμερα τίθεται και το θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών βέβαια. Αν χάσουμε κάποιον από αυτούς τους εταίρους καταλαβαίνετε ότι τίθεται σε κίνδυνο ολόκληρο το πρόγραμμα. Αλλά υπάρχουν και εσωτερικά προβλήματα τα οποία συζητάμε σε κάθε συνάντηση που έχουμε. Μια διαφορετική άποψη για το ενεργειακό μείγμα. Θέλουμε μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και στο μέλλον κάποιες χώρες μέλη μπορεί να είναι κατά της ε, σύνδεξης, τότε το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα δυσκολευτούν να δικαιολογήσουν τη χρηματοδότηση ενός τέτοιου προγράμματος. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Στο συζητάμε λοιπόν και αυτό. Σας ευχαριστώ για την εκθεσή σας. Ο κύριος Σαβανάτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με χαρά επισκέφθηκα το Καραντά. Ξεκαθαρίσαν στο μυαλό μου ιδέα πώ λειτουργεί το πείραμα. Είμαι πεπισμένο, Πρόεδρε, ότι θα σα ευχαριστούσα. ξέρετε ότι είσαι άνθρωπο των επιστημών, χημικό ε, και θα είσαστε ικανοποιημένο να βλέπετε αυτά που γίνονται εκεί. Εγώ είμαι από την Πάδοβα. Στην Πάδοβα γίνεται πειραματισμό για την πυρηνική σύνδεξη. Ε, RFX reverse uh, field experiment. Και από χρόνια, ήμουν δήμαρχος της Πάντοβα για πολλά χρόνια, και για χρόνια λοιπόν παρακολουθώ το πείραμα. Θέλω να σας διηγηθώ ε, κάτι ενδοτικά. Πριν από 30 χρόνια, ο καθηγητής Τζόρτζ Ροστάντο ήταν διευθυντής του προγράμματος φίλος μου. Του λέω, πότε θα φτάσουμε στη σύνδεξη Τζόρτζο, μου λέει. Σε 20 χρόνια θα φτάσουμε, μου λέγε. Μετά από 10 χρόνια περίπου, ρώτησα, Γιώργο, πότε θα φτάσουμε στην πυρηνική σύνδεξη. Έλεγε σε 30 χρόνια θα τα καταφέρουμε. Περνάνε άλλα χρόνια και ρωτάω, Γιώργο, πότε θα φτάσουμε στην πυρηνική σύνταξη. Μου λέει σε 40 χρόνια θα τα καταφέρουμε. <laughs> Κανονικά. Λοιπόν, είχα την επιβεβαίωση αυτή τη σειρά τη αυτή. Ξέρετε, αποκλίνουσε σε σειρά. Όσο περνάει ο χρόνο, τόσο πιο πολύ χρόνο χρειάζεται για να ολοκληρωθεί. Και κάπου ανησύχησα λίγο διότι το μηχάνημα που κατασκευάζουν δεν κάνει την πυρηνική σύνταξη που παράγει ενέργεια. Προσοχή. Αποδεικνύει ότι για μια περίοδο σημαντική, μεγάλη μπορούμε να έχουμε ελεγχόμενη σύνδεξη σε ένα περιβάλλον συγκεκριμένο που είναι το τόρο τόκαμακ. Αλλά δεν παράγει ενέργεια. Χρειάζεται άλλο μηχάνημα για να παράξει ενέργεια. Το ντέιμον θα αποκαλείται. Πού θα γίνει δεν ξέρω, πόσο θα κοστίσει δεν ξέρει κανείς. Αν υπάρχει πρόγραμμα όχι. Λοιπόν, κάνουμε ένα πείραμα για να δούμε αν μπορούμε μακροπρόθεσμα να διατηρήσουμε μια σύνδεξη δευτερίου και τριτίου. Το 2035 θα δούμε αν θα γίνει αυτό. Αλλά η σύνδεξη που παράγει η ενέργεια, σύμφωνα με αυτά που μου είπαν, χρειάζεται να περιμένουμε τον επόμενο αιώνα να γίνει αυτό. Λυπάμαι για σας, αλλά και για μένα, Πρόεδρε, έχω την εντύπωση ότι εκτός αν γίνει κάποιο θαύμα μέσω άλλης επιστήμης, δεν θα τα καταφέρουμε να τα δούμε τα υπέρ και τα κατά. Θα είμαι γρήγορος σε αυτό. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά υπέρ. Πρώτα απ' όλα η ποσότητα τεχνολογικής προόδου και παρεπόμενων ε, ανακαλύψεων για υλικά, για επικοινωνία, για μεταβίβαση στοιχείων κλπ. Είναι ενδιαφέρον αυτές εξελίξεις. Και όλος ο κόσμος συνεργάζεται και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Δίπλα στους ε, Ευρωπαίους με τους 45% έχουμε τις μεγάλες δυνάμεις και η Κορέα ακόμα είναι μέσα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, Ρωσία, όλοι είναι μέσα. Και αυτό είναι θετικό. Και είναι θέμα ειρηνικό, δηλαδή μαζεύεται ο κόσμο για να συζητήσει, να ψάξει να βρει με μεγάλη εναλλακτική. Αν κάποιο μου πει ότι αυτό θα σώσει τον πλανήτη από το φαινόμενο τη θέρμανση, δεν είναι στην ε, χρονική κλίμακα που συμβαίνει το φαινόμενο της αλλαγής του κλίματος. Εμείς κάνουμε ένα άλλο πείραμα και μετά θα δούμε αν θα φτιάξουμε το μηχάνημα. Μετά κάποιος πρέπει να φτιάξει ένα μηχάνημα που μπορεί να παράξει λογικό κόστος στην ενέργεια. Ε, και όλα αυτά δεν το βλέπω ε, να γίνεται γρήγορα όλα αυτά. Θετι... Αρνητικές στοιχές. Κάποια με έπληξε πολύ μεγάλο κόστος όπως υπενθυμίστηκε πρόσφατα τώρα εδώ ο χρόνος. Πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα που απαιτείται και ένα κάτι που από ό,τι κατάλαβα, λοιπόν, ε, ε, ε είμαστε κάπως ευαίσθητη θέση. Οι επιστήμονες ζωτάνε. γιατί είμαστε σε μια περιοχή που είναι κάπως ευαίσθητη. Ε, λέω εγώ, εσείς αποφασίσατε που θα κάνετε την εγκατάσταση που είναι ευαίσθητη ε, και αυτό με ανησυχεί κάπως η τοποθεσία. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι αυτή είναι ενδιαφέρουσα προοπτική είναι σαν το πρόγραμμα για να πάμε στον Άρη. Έχει πολλές πολλά θετικά αποτελέσματα παρεπόμενα, αλλά βλέπω ένα κοντινό ορίζοντα για να ωφεληθούμε από αυτή την ενέργεια, να έχουμε τελικά να αποκομίσουμε τα ωφέλη από την παραγωγή της ενέργειας. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραίες οι θέσεις σας, ήταν συναρπαστικότατες και πιστεύω ότι έπρεπε να είναι πραγματικά κάτι το πραγματικά ανευπροηγουμένου και χωρίς καμιά σχέση με την πραγματικότητα αυτό που είδατε θέλω να ενθαρρύνω και άλλους συναδέλφους γιατί όταν μίλησα με τον Γενικό Διευθυντή του ΙΤΕΡ συζητήσαμε τη δυνατότητα αυτή φυσικά είναι στη χώρα του είναι Γάλλος και οργάνωσε αυτή την επίσκεψη και συμφωνήσαμε ότι θα γίνει και μια άλλη επίσκεψη σε λίγες ε, Εβδομάδε και ίσω στην αρχή του επόμενου χρόνου θα γίνει άλλη μια επίσκεψη γιατί ήθελε να αποφύγει μια επίσκεψη 12-13 ατόμων από την Ήτρε. Καλύτερα πάνε 6 γιατί είναι πιο εύκολο. Θα οργανωθεί λοιπόν από την Κομισιόν μία ακόμα επίσκεψη και αν κάποιος θέλει να ε, ακούσει αυτά τα οποία είπατε, όλοι θα κινητοποιηθούν απάντες. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για τη συναρπαστική αυτή. Και ο κύριος Φρόιντ πάλι, Δέκα δευτερόλεπτα απλώς να σας πω, για αυτούς που ενδιαφέρονται σε αυτό το βίντεο, αλλά που δεν μπορώ να σας δείξω εδώ, για τεχνικούς λόγους, το βίντεο είναι στο διαδίκτυο, στο YouTube, με το όνομά μου, Eugen Freund, Ήτερ, μπορείτε να δείτε ότι μέσα σε δύο λεπτά παρουσιάζει αυτά τα οποία συζητήσαμε. Το βίντεο λοιπόν υπάρχει στο YouTube. Μετά από την επίσκεψή μου στο Ίτερ θα δω το βίντεο σου. Δεν θα το δω αντί να πάω εκεί πέρα. Θα πάω και θα το δω μετά. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Τρεις η ώρα επανερχόμεθα και αύριο βέβαια έχουμε τις ψηφοφορίες. Ευχαριστώ πολύ.